Mes chers collègues, bonjour. Venez prendre place, Monsieur Wim van de Kamp. Καλημέρα, καθίστε παρακαλώ. Θα ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας. Με τις ανακοινώσεις της Προέδρου σχετικά με τις αποφάσεις που έλαβαν οι συντονιστές. Έχετε λάβει και τα αντίγραφα. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις μέχρι τις 12.30 θα θεωρηθούν ως δεκτές. Ας περάσουμε τώρα στην ψηφοφορία. Ας ε, κάνουμε μια δοκιμαστική ψηφοφορία. Ένα τεστ λοιπόν. Για να δω Έχετε καλή διάθεση, ναι ή όχι. Για να δούμε ποιοι έχουν καλή διάθεση. Εγώ πάντως έχω. Είναι, έχουν ένα παραπάνω πράσινο, οπότε εγώ δεν θα ψηφίσω. Για δούμε η Επιτροπή τι θέση έχει. Τρεις δεν έχουν κέφια, βλέπω. Ένα, μία ψηφορία με ονομαστική κλίση για τον κύριο Τελίτσκα. Εντάξει. Αστείευαμε. Ξεκινάμε λοιπόν πολιτική συνοχή και θεματικό στόχο για την παραγωγή των βιώσιμων μεταφορών και την εξάλληψη των σημείων συμφόρηση στι υποδομέ των βασικών δικτύων. Την έκθεση του κυρίου Ζλωτόφσκι. Καλημέρα σα. Συμβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 21. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 28 υπέρ κατά Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 34. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές. Η ηλεκτρονική επαλήθευση άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται 34. Συνεχίζουμε. μεταστική 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 44β. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία. Α, θέλετε να απολυθέψουμε. Εντάξει. Άρχεται η ψηφοφορία για την 44β. Πέρας. Εγκρίνεται η 44β. Να με πιστεύεστε. 47 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 48 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 50 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 51 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 4 υπέρ Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 11. επέ. Κατά. Ο κύριος Βαντερκάμπ τι κάνει εκεί. Κύριε Μαρινέσκου, τους μπερδεύετε όλους. Πάμε πάλι. Για την 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Σημαστική 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Α, περνάμε στην τελική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας. Έγκρινεται. 35 ψήφοι. Υπέρ, 3 κατά, μία αποχή, συγχαρητήρια στον εισηγητή. Allez, nous continuons. Nous allons... Ας προχωρήσουμε λοιπόν να ψηφίσουμε τη διασφάλιση του ανταγωνισμού στον τομέα των αερομεταφορών. Έκθεση του κυρίου Μάρκους Πίπερ. Allez, nous commençons. Le compromis 1. Qui... Συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ογδόντα έξι υπέρ. Α, καταπίπτει, συγγνώμη. Η 74 εγκρίνεται αυτομάτως, επομένως η 86 καταπίπτει. Συμβαστική 2. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 102 τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται θα επαληθεύσουμε άρχεται πέρας Η τροπολογία 102 εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 106. 107 μάλλον. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται. Θέλετε να ελέγξουμε. Εντάξει, ας επαληθεύσουμε. Για την 107, άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται η 107. 108, υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 109, υπέρ. Κατά αποχές. Δεν ξέρω. Ας ελέγξουμε λοιπόν. Δεν ήταν σαφές. Πέρας. Για 109 λοιπόν. Πέρας λοιπόν. Εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 70 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έγκρινεται. Συμβαστική 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έγκρινεται. Συμβαστική 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 183. Υπέρ κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 184 υπέρ. Α, καταπίπτει. Και 185. Συμβαστική 9 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 10 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έγκρινεται. Συμβαστική 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έγκρινεται. Τροπολογία 170 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 179. Καταπίπτει. Το ξέρω, το ξέρω. Τροπολογία 181. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 186. Υπέρ κατά αποχές ας ελέγξουμε άρχεται πέρας Η ισοψηφία επομένω απορρίπτεται. Η 186. Συμβαστική 14 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 191 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται αυτή. Συμβαστική 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται και αυτή. Εκόν 31-32 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 239 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 240 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τρεις ταυτόσημες 241 έως 43 μια στιγμή Α, αυτές εκπίπτουν ή καταπίπτουν. Δεν ψηφίζονται. 244 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται, λέει η πρόεδρος, με κάποιο δισταγμό στη φωνή. Ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. 244. Πέρας. Α, να μην πιστεύεστε. Συνεχίζουμε. 244 λοιπόν απερίφθη. 245 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Α, προτιμάται η επαλήθευση. Αρχίζει. Τέλος. Απερίφθη. Πάλι καλά που το είδατε. Συνεχίζουμε. 246. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Οι επόμενες τρεις, 247 έως 249, εκπίπτουν. 33. Έκον. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Επαλήθευση ηλεκτρονικά. Ορίστε λοιπόν αρχίζει. Έκον 33. Πέρας. Έγκρινεται. Άρα λοιπόν να σηκώνετε καλά τα χέρια. Οι επόμενες τρεις, 250 έως 52, εκπίπτουν αυτές. Και προχωρούμε στην 253 και την 34 καθώς και τη 262. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές πάλι το αποτέλεσμα. Ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Τέλος. 26 υπέρ. Άρα εγκρίνεται. Συνεχίζουμε με την 263. Ψήφι υπέρ. 263. Με συγχωρείτε λέει πρώτος μια στιγμή. Η ΕΚΟΝ 34 εγκρίθηκε, άρα εκπίπτει. Πηγαίνουμε στην 254. 254 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Οι υπόλοιπε αυτές οι μεγάλη σειρά αυτή εκπίπτει επίση. 265 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική δέκατα. 82 το 82 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 285 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 289 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και αυτή. Ακολουθούν 3, 290 έως 92, αυτές εκπίπτουν. Και ακολουθεί, μια στιγμή, δύο ταυτόσημες, 293 και 94, ταυτόχρονα λοιπόν, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνονται, εγκρίνεται, εγκρίνονται οι δύο. 295 θέλετε επαλήθευση για την 293 και 4. Καλώς, αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνονται. 295 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 296, 7 και 8 εκπίπτουν και αυτές. Τροπολογία 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 299. Α, εκπίπτει αυτή, μάλιστα. Η 300 επίσης. 301 υπέρ. Κατά αποχές απόλυπτεται Συμβιβαστική 18 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία, με συγχωρείτε, 84 Α, ψηφίζεται, ψηφίζεται. 84 λοιπόν, υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται αυτή. Προτιμάται να γίνει επαλήθευση. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 16. Ψηφί υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα γιατί δεν σηκώνω όλοι καλά τα χέρια. Εσείς κύριε Πίπερ, ορίστε. Μιλώ για την 17. Ψηφίσαμε την 18, λέει ο κ. Πίπε. Όχι, όχι, όχι. 17. 17. Ας αρχίσουμε ξανά λοιπόν. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έκον 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έκον 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και έκον 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται και αυτή. Συμβαστική 19 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Εκόν 5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Έκον 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έκον 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έκον 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Έκον 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 30 έχει αποσυρθεί. Συμβαστική 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 41 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται έκον 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 21 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 52 έχει αποσυρθεί, 53 υπέρ, κατά, αποχές, δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα, ας επαληθεύσουμε, αρχίζει η ψηφοφορία 53. Πέρας. Δεν ήταν, προφανώς δεν ήταν σαφές το αποτέλεσμα. Άρα απορρίπτεται. Τροπολογία 55 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 13 εικόν 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 56 εκπίπτει 57 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 60 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται.

77 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές ψηφοφορία λοιπόν ηλεκτρονική αρχίζει πέρας η 77 εγκρίνεται 76 αυτή εκπίπτει. 80 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 85 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 61 εκπίπτει. 88 Έχετε ένσταση κατά της ψηφοφορίας κατά τμήματα. Όχι. Καλώς. Το πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Προχωρούμε τώρα στην ψήφιση του τελικού του σχεδίου. Αρχίζει. Τέλος. 28 ψηφί υπέρ, 9 κατά και 2 αποχές. Εγκρίνεται λοιπόν η έκθεση του κυρίου Πίπερ. Μην ε, φύγετε όμως και αμέσως εσείς κύριε Βαντεκάμπ θα ψηφίσουμε τώρα την διαπραγματευτική εντολή. Αρχίζει η ψηφοφορία. Έχει αρχίσει η ψηφοφορία. Κύριε Ανταπαντέλ, σας θυμίζω να ψηφίσετε. Πέρας. Εγκρίνεται λοιπόν με ψήφους 34 υπέρ κατά αποχές και καμιά αποχή. Η διαπραγματευτική εντολή λοιπόν έχει εγκριθεί. Προχωρούμε. Στο επόμενο θέμα της ημερησίας διατάξεως. Ξαναρχόμαστε στο πακέτο για την κινητικότητα και στην επιβολή τελών στα βαριά φορτηγά οχήματα κλπ. με την κυρία Ρεβόντα Λόν και άλλους συναδέλφους. Παρακαλώ, όσοι θέλετε να αποχωρήσετε, να το κάνετε ήσυχα. C'est mieux de laisser quelques secondes pour le... parce qu'il y a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 θα συνεχίσουμε με διαφορετική συζήτηση τώρα, αλλά πολύ σημαντική για το πακέτο που αφορά την κινητικότητα, συγκεκριμένα το πρώτο πακέτο κινητικότητας. Συγκεκριμένα έχουμε 2.309 τροπολογίες, 2.309 τροπολογίες που έχουν κατατεθεί, κάτι το οποίο δείχνει το μεγάλο ενδιαφέρον που έχει προκαλέσει αυτό το θέμα στην Επιτροπή μας. Οι συγητές και οι σκιώδεις, οι συγητές θα πρέπει να εργαστούν σκληρά ώστε να καταλήξουμε σε συμβαστικές τροπολογίες πριν από την ψηφοφορία στις 29 του Μάη. Καταλαβαίνω ότι δεν θα είναι εύκολο, αλλά νομίζω μπορούμε να επιδείξουμε μια συλλογική ευφυΐα και να τα καταφέρουμε. Από Οπότε συνάδελφοι, εύχομαι να έχουμε καρποφόρες συνεδρίες από σήμερα, ώστε να πετύχουμε τις απαραίτητες πλειοψηφίες για τους συμβασμούς. Θα ακούσουμε τους συναδέλφους για αυτό το ευρωσήμα και την περιβόητη οδηγία. Μετά θα ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά θα ζητήσω από τους εισηγητές να ολοκληρώσουν. Κυρία Ρεβονταλόν, έχετε το λόγο. Πολύ ευχαριστώ. Για την ημερομηνία της ψηφοφορίας 29 Μαΐου δεν είμαι σίγουρη. Είμαστε στο Στρασβούργο 29 Μαΐου. Πρόεδρος. 24 από ό,τι βλέπω προς το παρόν λέει πρόεδρος. Οπότε λάθος είπατε πρόεδρε προηγουμένως 29. Ναι, 24. 24 και μετά θα πάμε στην Ολομέλεια. Θα επανέλθουμε πάντως. Εντάξει, πολύ ωραία. Ξεκινάω λοιπόν. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί σκιώδες ηγητές, έχουν καταθεί πάρα πολλές τροπολογίες στο πλαίσιο αυτού του αριθμού του συναλλικού που αναφέρατε πρόεδρε. 483 για το συγκεκριμένο θέμα. Και αυτό δείχνει ακριβώς το ενδιαφέρον που έχει προκαλέσει αυτό το ζήτημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα τέλη. Δεν θα αναφερθώ σε όλες τις προτάσεις που περιλαμβάνουν οι τροπολογίες, αλλά σας αναφέρω τους κυριότερους προσανατολισμούς που αποκύπτουν. Θα ήθελα να διαπιστώσω καταρχάς ότι υπάρχει διακόπτη ομιλήτρια. Ξαναρχίζω γιατί Κάντε βασαρία. Θα πάμε λοιπόν προς σήματα και τέλη που έχουν να κάνουν με κύριο χαρακτηριστικό την απόσταση όσον αφορά την χρήση αυτών των υπηρεσιών. Κάποιοι θέλουν για το 2022 να μπει ένα τέλος όσον αφορά αυτά τα σήματα τελών, άλλοι επιθυμούν να υπάρχει διάκριση ε, σε σχέση με το βάρος των οχημάτων και νομίζω ότι υπάρχει επί της ουσίας μια συνένεση για να θέσουμε τέλος στο σύστημα των σημάτων τελών. Θα ακούσουμε στη συνέχεια ποια θα είναι η προθεσμία και νομίζω ότι θα πετύχουμε ένα σωστό συμβασμό στις τροπολογίες. Καταγράψαμε βεβαίω και τις απόψεις κάποιων βουλευτών που θέλουν να διατηρηθούν αυτά τα σήματα τελών. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι η πλειοψηφία των βουλευτών είναι έτοιμη να προχωρήσουν και να περιλάβουμε ε, και τα λαφρά οχήματα στο πεδίο εφαρμογή τη οδηγία. Μετά, για την αρχή του ΕΡΠΕΝ πληρώνει, θα πρέπει να σα πω ότι απογοητεύτηκα σχέση με το επίπεδο φιλοδοξία κάποιων συναδέλφων που έχουν καταθέσει τροπολογίε που θέλουν να επιβληθεί μια αρχή ανάλογα με την εκπομπή των ρήπων. Θεωρώ ότι η ε, εξωτερικοποίηση των εξωτερικών, του εξωτερικού κόστους σημαίνει ότι δεν θα είμαστε, σε θέση, θα είμαστε σε θέση να εφαρμόσουμε τις δεσμεύσεις μας για το περιβάλλον. Αυτή η οδηγία λοιπόν πρέπει να αποτελέσει ένα σημείο καμπής όσον αφορά την αρχή να πληρώνει. Πάντως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ούτως ή άλλως τα αποτελέσματα τα οποία θα έχουμε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Μετά, για την προσβασιμότητα των συστημάτων τηλεδιοδίων. Χαίρομαι που οι περισσότεροι Ευρωβουλευτέ έχουν καταθέσει τροπολογίε, οι οποίε ακριβώ ενισχύουν την εισηγησή μου για να λάβουμε υπόψη μα περισσότερο του κοινωνικο οικονομικού παράγοντε όσον αφορά τη διαβάθμιση των τελετιωδίων. Να πω επίση ότι έχω λάβει υπόψη μου τι ε, τροπολογίε των συναδέλφων σχετικά με τι ορεινέ περιοχέ, οι οποίε είναι ευαίσθητη σημασία για τι ε, δικέ μεταφορέ, Λαμβάνοντα υπόψη βεβαίω και ε, τι επιπτώσει που έχουν αυτά τα τέλη στην οικονομία και στου πολίτε αυτών των περιοχών. τέλο για τι συμβάσει παραχώρηση τη υπάρχουσα ε, που αφορούν όλε τι τωρινέ διατάξει. Βεβαίω θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μα την ισορροπία στι συμβάσει παραχώρηση. Όμω αυτέ οι συμβάσει θα πρέπει να είναι σε θέση να τροποποιηθούν και να προσαρμοστούν ανάλογα με το ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο. Να σα δώσω ένα παράδειγμα. Θα μπορούσαμε να ολοκληρώσουμε σε 10 χρόνια όσον αφορά τι διατάξει οι οποίε ισχύουν αυτή τη στιγμή στι περισσότερε ευρωπαϊκέ χώρε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ την εισηγήτρια Λαϊκή Πρόεδρο. Θα ξεκινήσουμε αμέσω τη συζήτηση. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Μπαρζόρ. Έχει το λόγο. Να ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, την Κριστίν Ρεβό για την θαυμάσια δουλειά της. Είχαμε δύο συναντήσεις ως σκιώδεις εισηγητές όπου συζητήσαμε το θέμα των ορισμών και κάποια άλλα κρίσιμα σημεία. Νομίζω ότι σε γενικές γραμμές είχαμε μια θαυμάσια συνεργασία και νομίζω ότι γνωρίζουμε όλοι ότι παραμένουν διάφορα δύσκολα σημεία που θα πρέπει να ρυθμίσουμε και τα οποία βέβαια θα προκαλέσουν σημαντικές συζητήσεις. Πάντως νομίζω ότι θέλουμε να είμαστε φιλόδοξοι σε σχέση με το Συμβούλιο το οποίο προσεγγίζει το θέμα αυτό με λιγότερο ενθουσιασμό θα έλεγα. Και δεν ξέρουμε ακριβώς ποιο τρόπο θα ακολουθήσουν διάφορες χώρες. Γι' αυτό ακριβώς θεωρούμε ότι θα ήταν καλό να έχουμε περιθώριο και χρόνο ώστε να επανέλθουμε στο θέμα. Γι' αυτό ακριβώς προτείνω να προχωρήσουμε θέτοντας σημαντικούς φιλόδοξους στόχους και θεωρώ ότι το θέμα θα μας απασχολήσει για πολύ καιρό. Το earmarking, το οποίο θα πρέπει να συζητήσουμε και το θέμα επίση του κόστους θα πρέπει να συζητηθούν στα πλαίσια του εξωτερικού κόστους. Και έχουμε και άλλο ένα σημαντικό ζήτημα που πρέπει να σχολιάσω. Λέμε ότι τα τέλη αυτά, τα διόδια είναι ακριβά και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και άλλους φόρους και τέλη τα οποία πρέπει να πληρώσει ο χρήστης. Νομίζω ότι αυτό όμως θα πρέπει να το τεκμηριώσει κανείς σωστά. ώστε να διατηρηθούν όλα αυτά σε ένα σωστό πλαίσιο. Το πρόβλημα τώρα με τις ε, συμβάσεις και αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει και να το συζητήσουμε σε βάθος και θα χρειαστεί να υπάρχει ασφαλεία δικαίου εδώ πέρα σε σχέση με τις ε, συμβάσεις παραχώρησης και θα πρέπει να δούμε κατά πόσο θα μπορέσουμε να προσαρμόσουμε την νομοθεσία για το μέλλον. Βεβαίω θα υπάρξουν ξαναλέω σημαντικέ αποκλήσει στις απόψεις μα, αλλά νομίζω ότι όσο έχει κάνει μέχρι τώρα η συγκήτρια μας βρίσκει σύμφωνους ιδιαίτερα όσον αφορά τις πιο σημαντικές αρχές. Ιδιαίτερα το να πληρώνουν αυτοί που χρησιμοποιούν αυτές τις υπηρεσίε. Και άλλες αρχές επίσης, βέβαια που ισχύουν και επίσης αναγνώριζεται από όλους. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Μπάρ. Ο κύριος Βαντελέν, έχετε το λόγο. Καλημέρα. Νομίζω ότι σε ό,τι αφορά τις αδρές γραμμές της αρχής ε, ο χρήστης πληρώνει, συμφωνούμε όλοι. Αλλά αλλά όντως ε, δεν ήταν όλα ομαλά μέχρι τώρα. Γιατί θέλω να υπενθυμίσω στους αδέλφους γιατί ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη συζήτηση για, για τα τέλη κυκλοφορίας και χρήση του δικού δικτύου δηλαδή. Ξεκίνησε επειδή αρχικά θέλαμε λιγότερα βαρέα οχήματα στο δικό δίκτυο γιατί αυτό τα βαρέα οχήματα ε, δημιουργούν φθορέα στο οδικό δίκτυο. Αλλά επειδή θέλαμε να βρούμε άλλους τρόπους μεταφοράς πιο φιλικούς προς το περιβάλλον. Αυτό το σημείο κίνησης, από ό,τι βλέπω, αποδυναμώνεται, κυρία Πρόεδρε. Η συζήτηση που κάνουμε αυτή τη στιγμή μεταξύ των σκιωδών εισηγητών μου δείχνει ότι κάποιοι λένε επιτέλους μπορούμε να προχωρήσουμε σε έναν ευρωπαϊκό φόρο, για να μην μιλήσω για ευρωπαϊκό φορολογικό παράδεισο για κάποιους. Εγώ σίγουρα δεν είμαι πέρα αυτής της προσέγγισης. Αλλά και άλλοι συνάδελφοι θέλουν ε, επιτέλους να ζήσουν το μεγάλο όνειρο, τη, τη μεγάλη τους αγάπη, το τις ευδρομικές μεταφορές, να τις ε, βάλουν στο θρόνο λοιπόν και να εκθρονίσουν το, τις οδικές μεταφορές. Νομίζω ότι προτρέχουμε, ειδικά σε ό,τι αφορά τα στοιχεία αυτά. Επιπλέον, Πρόεδρε, πρέπει να δηλώσω την απογοήτευσή μου σε σχέση με ορισμένες πολιτικές ομάδες για, τις, ε, για τους τρόπους μεταφοράς που είναι φιλικοί προς το περιβάλλον. Και πιο συγκεκριμένα θέλω να αναφερθώ και στα λεωφορεία και στα μοτοποδήλατα Πρόκειται για τρόπους μεταφοράς που είναι φιλικοί προς το περιβάλλον. και σίγουρα ε, καταπολεμούν και τη συμφόρηση, αλλά άλλοι συνάδελφοι λένε όχι και τα λεωφορεία και τα μοτοποδήλατα θα πρέπει να μπουν ε, σε αυτή την κατηγορία. Αλλά πραγματικά μου διαφεύγει η επιχειρηματολογία αυτή. Και ιδίω ό,τι αφορά τι πολιτικέ ομάδε που ε, επιμένουν να μπει στη συζήτηση και το λεωφορείο. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω. Και ήδη ε, και στη συζήτηση των σκιωδών το έχω επισημάνει ότι αυτό θα είναι πρόβλημα για μένα. Τέλος, κύριε Πρόεδρε. Τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα. Η ποιότητα είναι το πιο σημαντικό και όχι το χρονοδιάγραμμα. Γιατί κάποιοι έτσι προσπαθούν ε, να μας εκβιάσουν, άντε, στα γρήγορα, μην καθυστερούμε. Για μένα είναι ένα από τα πλέον σημαντικά ζητήματα στις μεταφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, το πιο σημαντικό είναι η ποιότητα. Αναφέρθηκε η προθεσμία της 24ης Μαΐου. Ε, για το ECR αυτή η ημερομηνία δεν μπορεί να λειτουργήσει, γιατί εγώ είμαι... Ε, έχουμε τις, ε, τα study days μας στο Ρότερνταμ και θα μιλήσουμε και για προγράμματα που αφορούν τις μεταφορές, θα μιλήσουμε και με προσώπους των λιμένων, της τοπικής αυτοδιοίκησης, οπότε θα ήθελα να το αναβάλουμε για αργότερα. Γιατί αυτό πραγματικά θα ήταν πρόβλημα από πλευρά ε, συντηρητικών και μεταρρυθμιστών. Από πλευρά παρουσία μα δηλαδή. Λοιπόν, είμαστε καθοδόν, είναι δύσκολο ο δρόμος. Ανέφερα ορισμένα ζητηματάκια που έχω εντοπίσει εγώ. Θα συνεχίσουμε τη συζήτηση με του συναδέλφους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Βαντελέν. Η 24η Μαΐου έχει τεθεί όχι για να μην ισχύσει, αλλά για να γίνουν όλα αυτά που θέλουμε. Δηλαδή να υφηθήσουμε το πρώτο πακέτο την πρώτη μέρα. Το πρώτο πακέτο λοιπόν καταρχάς και μετά ξαναλέω θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή όλα αυτά τα θέματα και τα σημεία που αφορούν το πρώτο πακέτο. Ο κ. Δρικέ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τη θαυμάσια εισηγησή του. Συμμεριζόμαστε το γενικό στόχο της εισηγησής Έχουμε την αρχή ο... Έχουμε την Και μέχρι τώρα είχαμε ένα θελοντικό πλαίσιο εφαρμογής για αυτές τις αρχές. Τώρα για το κατά πόσο αυτά τα σήματα τελών θα εξαφανιστούν ή όχι, δεν ξέρω. Υπάρχει ένα θέμα πάντως ε, συνέπειας, ομοιογένειας, διαφάνειας σε όλη την Ευρώπη νομίζω. Και όπως είπε προηγουμένως και ο Τζόρς, το earmarking μου φαίνεται σημαντικό. Είναι αλήθεια θα είναι δύσκολη μάχη με το Συμβούλιο. Παρ' όλα αυτά υπάρχει μια ηθική λογική εδώ σε αυτή τη, διά, διάταξη σε σχέση με την αποδοχή της από αυτούς που υπόκειται σε αυτό το τέλος. Δηλαδή το earmarking έχει γενική ισχύ. Πάντως το θέμα είναι νομίζω αρκετά δύσκολο γιατί αφορά τα οικονομικά. Αφαιρθήκαμε και στις συμβάσεις παραχώρησης. Διάβασα τον τύπο και ανησύχησα να σας πω την αλήθεια γιατί νομίζω δεν καταλαβαίνουν ε, καλά αυτό που έχουμε προτείνει. Τώρα για την ασφάλεια δικαίου έχουμε τις οδηγίες, πρέπει να τηρηθούν και θα πρέπει να είμαστε τουλάχιστον συνεπείς με τους εαυτούς μας. Πάντως, αυτές οι συμβάσεις παραχώρησης είναι συμβάσεις απόσβεσης. Δεν μπορούμε να επαναφορολογήσουμε αυτή την ε, απόσβεση του κόστους. Θα πρέπει αυτές οι συμβάσεις παραχώρησης να μην αλλάζουν ριζικά και θα πρέπει να μπουν στο γενικό πλαίσιο διατάξεων στον έχουμε ακριβώς ασφάλεια δικαίου. Εγώ θα ήθελα επίσης να καθορίσουμε και το γενικότερο πλαίσιο αυτού του εθνικού φορολογικού πλαισίου που αφορά τα τέλη και τα διόδια. Μετά και για τις ε, τοπικές αρχές και αυτές θα πρέπει να είναι σε θέση να κάνουν ε, μια διαφοροποιημένη εφαρμογή, όπως ακριβώς νομίζω θα ισχύει σε διάφορες χώρες, θα έχουμε περιφερειακή εφαρμογή, τοπική εφαρμογή και θα είναι λοιπόν απαραίτητο οι συλλογικές, οι συλλογικότητες οι τοπικές να είναι σε θέση να συμμετάσχουν κατάλληλα. Επίσης, για τα ιστορικά οχήματα, αυτό το σημαντικό κομμάτι της κληρονομιάς νομίζω δεν θα έχουν δυνατότητα να κυκλοφορήσουν. Θα πρέπει να δούμε και τον ιστορικό τους χαρακτήρα και το πώς εντάσσονται στο συνολικό πολιτιστικό πλαίσιο. Αυτά από μένα. Ελπίζω πάντως να βρεθούν πλειοψηφίες και συμβασμοί και μάλιστα, όπω είπε και ο, Ζόρ, τη στιγμή που η συζήτηση με το Συμβούλιο δεν θα είναι και τόσο εύκολη. Και Ρικέ, σα ενδιαφέρει πολύ η DS, η Citroën DS του Charles de γι' αυτό φαίνεται. Ναι, αλλά είχε υπάρχει κάποια ζημιά νομίζω, σε κάποια τρομοκρατική ενέργεια. Παρακαλώ, επόμενο ομιλητή. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ και την εισηγήτρια και για το σχέδιο, αλλά και για την και την καλή συνεργασία που είχαμε μαζί της, γιατί το θέμα είναι περίπλοκο. Έχουμε λοιπόν μια κατάσταση όπου πράξεις και έργα αποκλίνουν πολύ στην Ευρώπη. Δηλαδή αφάνταστο χάος. Είμαι 14 χρόνια ευρωβουλευτής. Η αρχή, ο χρήστης πληρώνει, ο ρηπαίνων πληρώνει, ε, Θεμητό ανταγωνισμό. Σε αυτά συμφωνούν όλοι. Απολύτως. Όταν όμως πρόκειται να τα εφαρμόσουν στην πράξη, όταν λέει κανεί, κοιτάξτε να εδώ ο, ο, είναι αθέμητο. Α, τότε όλοι κάνουν ότι κοιτούν αλλού. Φανταστείτε, αν είμαστε έτσι εμεί, τότε πώς θα αντιδράσει το Συμβούλιο Υπουργών. Και δεν άρχισε η υπόθεση με τα διόδια στους δρόμους, αλλά με τα διόδια στα τρένα, στους σιδηροδρόμους, όπου δεν υπήρξε δεσμευτική νέα ρύθμιση έχουν επιβάλει διόδια στις ε, μηχανές έλξιος ανά χιλιόμετρο που διανύουν. Πολύ όμως προτιμότερος ο σιδηρόδρομος από τον αυτοκινητόδρομο, το γνωρίζετε από άποψη ρηπάνσεως, εάν ο σιδηρόδρομος, μάλλον εάν ο αυτοκινητόδρομος ήταν φιλικός στο περιβάλλον, θα έλεγα εντάξει, να μην βάλουμε διόδια. Αλλά συμβαίνει το αντίθετο. Εμεί βλέπουμε διαρκώ την Ευρωπαϊκή Ένωση και τι χώρε μέλη να υποστηρίζουν, να επιδοτούν, να ευνοούν τι μεταφορέ που είναι οι πιο ρηπογόνε και να επιβάλλουν ποινέ στην ουσία στους λιγότερο ρηπογόνου τρόπου μεταφορών όπω είναι ο σιδηρόδρομο. Ό,τι στόχου και να διατυπώνουμε για την προστασία του κλίματο, δεν θα τα καταφέρουμε ποτά, ποτέ διότι οι μεταφορές είναι κατά 40% συνολικά υπεύθυνε για τη ρήπανση και 70% μέσα στις πόλεις. Είμαι πεπισμένος ότι μπορούμε να επιτύχουμε για κινητικότητα και να προστατεύσουμε και το κλίμα, αλλά με σωστά μέτρα. Και ούτε χρειάζεται να κάνουμε επινόηση του τροχού εκ νέου. Οι Ελβετοί υπάρχουν οι οποίοι μας δείχνουν το σωστό δρόμο. Διόδια στα φορτηγά αυτοκίνητα που αρχικά άρχισε για να χρηματοδοτηθεί η ε, σύραγγα του Γκοτάρ, και ισχύει πλέον σε όλου τους δρόμους για όλα τα φορτηγά αυτοκίνητα άνω των 3,5 τόνων. Και επομένως δεν μεταφέρουν τα φορτία από τα μεγάλα φορτηγά που επιβαρύνονται στα μικρά φορτηγά, τα οποία επιβαρύνονται λιγότερο. Οι Ελβετοί λοιπόν είναι έξυπνοι και εμεί είμαστε χαζοί και δεν μπορούμε να μιμηθούμε το παράδειγμά του. Αυτή είναι η κατεύθυνση που πρέπει να κινηθούμε. Ευχαριστώ την Ελβετία Πιθανώ είναι τόσο Ευρωπαίοι στο πνεύμα, μόνο και μόνο επειδή δεν είναι μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι χρειάζεται λοιπόν τώρα. Η μελέτη δεν περιλαμβάνει τα πάντα. Θα πρέπει να μπουν μέσα και τα ατυχήματα και ούτω καθεξής. Το κάθε αυτοκίνητο που κυκλοφορεί στην Ευρώπη επιδοτείται από χρήματα των φορολογουμένων με 1.600 ευρώ το χρόνο. Εγώ εδώ 40 χρόνια δεν έχω αυτοκίνητο και όμως έχω πληρώσει χιλιάδες ευρώ σε φόρους για τα αυτοκίνητα. Δεύτερο, η συγχρηματοδότηση. Με την Επιτροπή Μεταφορών, έχει καιρό που είχαμε πάει στην Ισπανία. Και κινηθήκαμε με το λεωφορείο πάνω σε ένα θαυμάσιο αυτοκινητόδρομο που είχε συγχρηματοδοτηθεί και σε πολύ ψηλό ποσοστό από την Ευρωπαϊκή Ένωση Βεβαίω όλοι αναμέναμε να υπάρχει πολύ μεγάλη κυκλοφορία. Κάθε μισή ώρα περνούσε ένα φορτηγό. Κοιτάξαμε μετά και τον διπλανό επαρχιακό δρόμο, τα φορτηγά το ένα πίσω από το άλλο. Γιατί, Γιατί στον επαρχιακό δρόμο δεν πληρώναν διόδια. Ενώ στο αυτοκινητόδρομο ναι. Είμαστε τρελοί. Επενδύουμε δισεκατομμύρια και βάζουμε συνθήκε πλαίσια που τελικώ οι υποδομέ αυτέ δεν χρησιμοποιούνται. Κανένα ιδιώτη δεν θα πέταγε τα λεφτά του έτσι από το παράθυρο. Εμείς όμως το κάνουμε στην Ευρώπη με ευρωπαϊκά χρήματα. Γι' αυτό λέμε εμείς καθαρά. Τα διόδια θα πρέπει να ισχύουν σε όλους τους δρόμους, ώστε να μην υπάρχει αυτή η μετατόπιση. Ευρωπαϊκά χρήματα δεν θα πρέπει να δαπανώνται για δρόμους εφόσον αυτοί έχουν διόδια. Δεν είναι δυνατόν με τα χρήματα που εισπράττονται σε κάποιες χώρες από τα διόδια να χρησιμοποιούνται μετά για δρόμους αλλού που δεν πληρώνουν διόδια. Όλα αυτά είναι αθέμητο ανταγωνισμός. Γι' αυτό και χρειαζόμαστε διόδια που να είναι πανευρωπαϊκά, δεσμευτικά για όλους, όπως γίνεται με τον σιδηρόδρομο, χρειαζόμαστε ελάχιστα ποσοστά, ελάχιστα ποσά μάλλον, ελάχιστα όρια των διοδίων, όπως γίνεται και στο σιδηρόδρομο άλλωστε. Κάπου είναι πολύ ψηλά τα διόδια για τα επιβατικά αυτοκίνητα, κάπου για τα φορτηγά. Πρέπει να τα εννοιοποιηθούν όλα αυτά. Όλα αυτά πρέπει να περιληφθούν και μόνο έτσι μπορεί να εξασφαλιστεί η κινητικότητα αλλά και να προστατευτεί το περιβάλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, συναδελφοί, καταρχάς να ευχαριστήσω την Κριστίν και τη θαυμάσια ομάδα σας. Ξέρω ότι ήδη κάνατε θαυμάσια δουλειά με τον τεράστιο αριθμό τροπολογιών και νομίζω ότι με μια καλή συνεργασία θα μπορούσαμε να βρούμε κάποιες λύσεις. Θα αναζητήσουμε λοιπόν λύσεις και, όχι... και θα επικεντρωθούμε στα προβλήματα. Γιατί τότε παραβλέπουμε τις λύσεις. Νομίζω ότι η βασική αρχή ο χρήστη πληρώνει, ο Ιρπιόν πληρώνει, νομίζω είναι ξεκάθαρη, τουλάχιστον για μας. Αλλά υπάρχουν ακόμα ζητήματα, όπως ας πούμε σχέση με τις δημόσιες μεταφορές και το πώς το στηρίζουμε αυτό. Δηλαδή, για να βελτιώσουμε τα πράγματα σχέση με σήμερα και πώς συνεργαζόμαστε με τις διάφορες περιφέρειες, σε αντίθεση δηλαδή με αστικές περιοχές ή άλλες περιοχές όπου έχουμε λιγότερη, λιγότερα χήματα που κυκλοφορούν, πιο αεροκατοικημένες, πιο πυκνοκατοικημένες. Υπάρχουν λοιπόν διαφορές και το θέμα για τις χώρες ε, μέλη είναι το πώς ακριβώς θα αναζητήσουμε και θα βρούμε ευέλικτες λύσεις για διάφορες ε, περιοχές και για διάφορες χώρες. Νομίζω ότι αν έχουμε ένα ευέλικτο, ευφυές και ανοιχτό σύστημα, όπου θα μπορέσουμε ακριβώς να μοιραστούμε και τα σημαντικά δεδομένα, τότε μπορούμε να βρούμε και λύσεις οι οποίες θα είναι καλύτερες για τις ε, χώρες από το να πούμε ότι θα έχουμε μια ενιαία λύση για όλους. Αν κάνουμε εξαιρέσεις, τότε θα πρέπει να τις εξετάσουμε σοβαρά και θα πρέπει να είμαστε λογικοί. Αλλά αυτό που κάνουμε συνήθως όταν μιλάμε για μετακινήσεις με λεωφορεία, ποδήλατα, ιδιωτικά οχήματα κτλ. Θα πρέπει να έχουμε πάντοτε κατά νου τις ε, πολυτροπικές μεταφορές και το πώς θα μπορούσαν να λειτουργήσουν σωστά αυτές. Νομίζω ότι θα πρέπει με τις δημόσιες μεταφορές να δούμε ακριβώς πώς θα κατανεμηθούν. Γιατί βλέπουμε ας πούμε να γίνεται μετακινήσεις ενός αυτοκινήτου με ένα άτομο μέσα και πάνε στην, έχουν τους ίδιους προορισμούς. Οπότε μπορούμε να προωθήσουμε ας πούμε το carpooling Το ίδιο και αλλού και σε άλλε περιπτώσει. Πάντω κάπω με ανησυχεί αυτό το πώ θα συνδέσουμε το θέμα τη φορολόγηση που προβάλλεται στις χώρες μέλη σε σχέση με τις μεταφορές και το πώς θα συνδέουμε όλα αυτά με τρόπο ευφυή με το ευρωσήμα τελών. Με ανησυχεί αυτό. Γιατί συνήθω τσακωνόμαστε με τις χώρε μέλη σε σχέση με την υπάρχουσα φορολόγηση των ε, μεταφορών. Πάντως, το μήνυμα από αυτές τις πάνω από 2.000 τροπολογίες είναι ότι είχαμε ένα χειμώνα κάπως παράδοξο στην Ευρώπη και όταν είπαμε ότι θα πρέπει να επενδύσουμε στο ευρωσήμα τελών για την ασφάλεια των μεταφορών ακριβώς και για να διασφαλίσουμε και τους χώρους στάθμευσης και τα τότε θα πρέπει να δούμε ακριβώς πώς θα είναι ασφαλή αυτά τα σημεία στάθμευσης για όλους, υπό ασφαλείς ηθίκες δηλαδή, καθόλου όλη τη διάρκεια του χρόνου, έτσι, και υπό διαφορετικές καιρικές συνθήκες. Καταρχάς λοιπόν θα πρέπει να αλλάξουμε την οτροπία μας και εδώ στην Επιτροπή μας και στην ομάδα μας για το Ευρωσήμα Τελών. Γιατί αν παραμένουμε προσυλλομένοι στην υποστήριξη ας πούμε, μιας και μόνο ιδέας, τότε θα είναι δύσκολο η Κριστίν να βρει συμβασμούς με την υπόλοιπη ομάδα. Αν όμως είμαστε ανοιχτοί, δεκτικοί και έχουμε υπόψη μας τους απότερους στόχους, τότε με σωστή συνεργασία θα βρούμε λύσεις. Για χάρη λοιπόν του Γιέντς Νίλσον θα πω κάτι στα σουηδικά. Θα πω λοιπόν. Θα πρέπει να δίνουμε μάχη ώστε να καταφέρουμε να είμαστε οι καλύτεροι σε αυτή την περίπτωση για αυτά που αφορούν βέβαια το Ευρωπαϊκό Συμματελόν. Με πολύ αγάπη από μένα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε που κλείσατε και με μία μνήα στο συνάδελφό μας Γιάννης Νέλσον. Κυρία Αγιούτο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Καταρχάς να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τη θαυμάσια δουλειά που έκανε και για την ε, δυνατότητά της να διασφαλίσει τους πυλώνες που έχουν ε, στηρίξει αυτή την πρόταση της Κομισιόν πάνω στην οποία δουλεύουμε. Οπότε στηρίζω και την αρχική πρόταση της Κομισιόν αλλά και την έκθεση της εισηγήτριας. Ιδιαίτερα θα πρέπει να κοιτάξουμε τη μετάβαση από τα τέλη που αφορούν χρόνο σε τέλη που αφορούν την απόσταση. Αυτό είναι το βασικό στοιχείο. Έχουμε και δύο σημαντικού παράγοντες. Καταρχάς, ο ένας αφορά τη σημασία του εξωτερικού κόστους, κόστους που αφορά τη συμφόρηση, αυτά θα πρέπει να επανενταχθούν στο σύστημα των μεταφορών. Οπότε για μας αυτό είναι βασικό και νομίζω ότι θα εμπλουτίσει τον το των υποδομών που σε κάποιες περιοχές των χωρών μελών υστερούν. Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα αφορά τη διαφάνεια. Τη διαφάνεια σε σχέση με τις επενδύσεις που έχουν γίνει και με την κατάλληλη διαφάνεια που θα πρέπει να δίδεται προς τους χρήστες όσον αφορά τα αποτελέσματα και της οδικής ασφάλειας αλλά και τα αποτελέσματα για το περιβάλλον και την υγεία και τις επιπτώσεις. Δηλαδή οι επενδύσεις που γίνονται θα πρέπει να είναι αντιληπτές από τους πολίτες άμεσα σε σχέση με τα θετικά τους αποτελέσματα. Διαφάνεια επίσης σε σχέση με τις αναφορές στο report των χρωμελών. Τώρα για τις δεσμεύσεις, μάλλον συγγνώμη για, τις, ε, για τους συμβασμούς, είμαστε θετικοί για την επέκταση και σε άλλα μέσα. Για το δευτερόγον τώρα δίκτυο όμως έχουμε κάποιες αμφιβολίες θα πρέπει νομίζω να αξιολογήσουμε σωστά και τον οικονομικό αντίκτυπο, ιδιαίτερα όσον αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις των μεταφορών, δηλαδή αν επεκταθούμε όσον αφορά τα τέλη και τα διόδια και στα δευτερεύοντα δίκτυα. Τώρα για τους χώρους στάθμευσης νομίζω ότι είναι σωστό να επενδύσουμε στην δημιουργία αυτών των χώρων στάθμευσης που θα είναι ασφαλείς και θα μπορούν να διασφαλίσουν και σωστές κοινωνικές συνθήκες στους ε, μπλεκόμενους οδηγούς, αυτοκινητιστές κτλ. Επίσης, δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε θαυμάσιους χώρους στάθμευσης, οι οποίοι από πλευρά ε, κόστους δεν θα είναι προσβάσιμοι, δηλαδή δεν θα επιλεχθούν ποτέ, ιδιαίτερα από τις ε, μικρές επιχειρήσεις επιμελητίας. Και τέλος, όπως είπαμε, συμφωνούμε και με το earmarking γενικά και στους συμβασμούς, πάντοτε στα πλαίσια της διαφάνειας και συμφωνούμε απόλυτα και με την πρόταση που υποβάλλεται για, το reporting. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Θα δώσουμε το, το λόγο στους υπόλοιπους συναδέλφους. Κύριε Κόρη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και την αγαπητή Κριστίν, ο κύριος Κοχ. Τώρα έχω το εξής. Πρώτον, το κόστος που προκαλούν οι εχμές κυκλοφορίας. Επιβαρύνει τους ε, χρήστες ήδη. Άρα να αυξηθούν τα διόδια πάλι θα επιβαρύνει τους χρήστες. Να φύγουν τα διόδια από την οδηγία αυτή. Τώρα να τα διαγράψουμε σε αυτήν την αναθεώρηση. σε κανένα δεν αρέσει να κάθεται μέσα σε εχμές και να πληρώνει κιόλα και να δαπανά το χρόνο του και το καυσιμό του και τα νεύρα του. Δεύτερο, χρειαζόμαστε δεσμευτική πρόβλεψη του στόχου που θα χρησιμοποιούνται τα χρήματα από τα διόδια για την βελτίωση των αποδομών, την εγγύηση της ασφάλειας των υποδομών και της βιωσιμότητάς τους. Τρίτο, διόδια τα οποία να υπολογίζονται διανιόμενη απόσταση. Μόνο αυτά είναι δίκαια. Διόδια στη βάση του χρόνου είναι ακατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν τα χρήματα από την ίσπραξή τους για την ασφάλεια των υποδομών. Συστήματα διοδίων που βασίζονται στον υπολογισμό του χρόνου πρέπει σταδιακά να πάψουν να λειτουργούν. Και τελευταίο, δεν μου αρέσουν πολύ οι εξαιρέσει. Όμω υπάρχουν κάποιε εξαιρέσει που είναι σκόπιμε. Και μια σημαντική θα ήταν να δοθεί η δυνατότητα στι χώρε μέλη να απαλλάξουν τα ιστορικά οχήματα που εν τέλει είναι και κληρονομικό αγαθό τη πολιτιστική μα κληρονομιά. Να τα εξαιρέσουν λοιπόν από την επιβολή διοδίων. Ο κύριο Βαν Κάμπ. Κυρία Πρόεδρε, σα ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την Κριστίν για την πολύ καλή αυτή ε, έκθεση. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς εδώ. Πρέπει κάπως να πρασινίσουμε εντό εισαγωγικών τις οδικές μεταφορές. Και συμφωνώ με τον κύριο Κράμερ. Πολλά έχουμε πει λοιπόν για την οικολογική διάσταση στις οδικές μεταφορές, όμως έχει έρθει η ώρα, πιστεύω, ε, πραγματικά να δείξουμε τι μπορούμε να κάνουμε σε Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω όμως ότι η κυρία εισηγήτρια σε ορισμένα σημεία ε, κάνει λάθος επιλογές. Ξεκινώ με το εξής ερώτημα. Ανάπτυξη της υπαίθρου και οδικές μεταφορές μεταξύ δύο χωριών, για παράδειγμα, στην υπαίθρο της Γαλλίας. Δεν γίνεται τώρα να βάλουμε διόδια εκεί. Κάποιε φορέ έχω την εντύπωση ότι είναι σαν να μένουμε όλοι στις πόλεις. Ίσως μένει συγγήτρια σε πόλη και έτσι είναι πιο εύκολο να ε, χρησιμοποιούμε όλη λεωφορεία και ε, Όμω Όμως τα πράγματα αλλάζουν. Δεν μπορούμε να επιβάλλουμε φόρους ε, στην Ήπεθρο. Γιατί έτσι καλώς έχει μειωθεί ο πληθυσμό σε αυτέ τι περιοχέ για παράδειγμα, στην Bundesstraße και σε τέτοια περιφερειακά οδικά δίκτυα, καταλαβαίνω ότι για να μειώσουμε ε, τη συμφόρηση βάζουμε διόδια. Γιατί αν όλοι πάνε από, το εθνικό δίκτυο στην Bundesstraße, τότε απλώς μετατοπίζουμε το πρόβλημα. Όμως, ως Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα διαφωνούμε με την φορολόγηση της υπαίθρου. Το ίδιο είπε ο συνάδελφος για τα τέλη συμφόρησης που είπε ο κύριος Κόχ. Αν πούμε ότι ε, προσδιορίζεται με βάση την απόσταση και με βάση τις εκπομπές υψηλίου του άνθρακα, τότε νομίζω ότι κάνουμε αρκετά. Και δεν θα αφήσουμε τους φίλους μας από την DHL και να πληρώσουν διόδια και να κάθονται και στην κίνηση. Τώρα για το earmarking. Ε, διαφωνώ εδώ με τον αγαπητό συνάδελφο Κοχ ε, διαφωνώ με το earmarking. Νομίζω ότι είναι επικίνδυνη οδός το earmarking από τεχνικής άποψης. Ε, για να σας αναφέρω την υποδοχή των ετούντων άσυλων. Δεν μπορούμε να πούμε, ας πούμε, όταν έχουμε τέτοιου είδους κρίσεις ότι δεν γίνεται γιατί αυτά τα χρήματα τα έχουμε αναθέσει και έχουμε κάνει earmarking για τα διόδια. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Τώρα για τους ε, κινητήρες καταλαβαίνω ότι υπάρχει ε, ιδιωτικό συμφέρον. Ο κύριος Βαντάλ λοιπόν το είπε πάρα πολύ ωραία και συμφωνώ. Ακούω σοβαρά μηνύματα από το Συμβούλιο ότι θέλουμε να θέσουμε σε ισχύ ε, την πρόταση αυτή σε περίπου 20 χρόνια. Μα δεν έχει κανένα νόημα. Ελπίζω λοιπόν η εισηγήτρια ε, να φέρει πιο κοντά στο παρόν ε, την θέση σε ισχύ γιατί καθυστερούμε ιδιαίτερως. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη δική μας λήψη αποφάσεων, με κάθε σεβασμό προς τον Πέτερ Βαντάλα, εγώ, εντάξει, μπορεί και να παντρευτώ στις 24 Μαΐου, ούτε εγώ μπορώ να έρθω να ψηφίσω. Είναι επικίνδυνη αυτή η προσέγγιση. Και σα στηρίζω κυρία Πρόεδρε να κάνουμε την ψηφοφορία στι 24 Μαΐου γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να λειτουργήσει, πρέπει να δουλέψουμε, γιατί όλο μιλάμε. Ζούμε σε μια φούσκα που σε, από κάποιες απόψεις δεν έχει καμία σχέση με την κοινωνία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Βαντρεκάμπ. Ε, το μόνο που εγώ κρατάω είναι ότι παντρεύεστε και δεν μας έχετε καλέσει. Στις 24 ό,τι και να έχετε να κάνετε, ε, πρέπει να έρθετε εδώ στην ψηφοφορία. Ο κύριος Φαγκρίνη έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ε, για τον κύριο Κοχ, είπατε για την πολιτιστική κληρονομιά, τα λεγόμενα οχήματα old timers. Ξέρετε ότι και εγώ τα αγαπώ, αυτά τα παλαιά αυτοκίνητα, τις αντίκες. Έχω ένα ε, παλιό Volvo το 89 με πάνω από 100.000 ε, χιλιόμετρα, αλλά μια χαρά πηγαίνει. Δεν χρειάζεται να παράξουμε ένα καινούριο όχημα για να το αντικαταστήσει. Οπότε συμφωνώ κύριε Κόχ. Αυτό είναι καλό για το μέλλον. Μετά, δεν νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει ε, να επιβάλλει τέλη για την χρήση των υποδομών. Αυτό είναι εθνική ερμοδιότητα κατά τη γνώμη μας. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες σε εθνικό επίπεδο. Για παράδειγμα, έχουμε τα δάση στη Σουηδία που ήταν πολύ δύσκολο λόγω των δασών να ε, φτιάξουμε το συνδρομικό δίκτυο. Δεν έχουμε δώσει χρήματα για τις υποδομές και είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο να μπει, να πάρει κανείς το τρένο στη Σουηδία γιατί κανείς δεν ξέρει πότε και πού θα φτάσει. Οπότε η καλύτερη ελεκτική λύση είναι τα ε, αυτοκίνητα και τα μεγαλύτερα βαρέα οχήματα, αυτά είναι η καλύτερη επένδυση για το περιβάλλον. Γιατί όταν έχουμε μεγάλε αποστάσει, πρέπει να ε, είμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε και μεγάλο φορτίο. Και το μεγαλύτερο κέρδος για το περιβάλλον είναι η βελτιστοποίηση των μεταφορών. Έτσι έχουμε καλύτερες αποδόσεις, καλύτερες από ό,τι αν επιβάλλουμε τέλη. Δεν ξέρουμε τι γίνεται με αυτά τα τέλη, τα διόδια. Ε, τα εθνικά τέλη καυσίμων θέλει τώρα να τα πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ως ίδιο πόρο. Αυτό προκύπτει από τις προτάσεις του κυρίου Έτιγκερ. Έχουμε πολύ ιδιαίτερες ε, συνθήκες στη Σουηδία. Η μεγαλύτερη περιβαλλοντική ανάγκη συνδέεται με τα λεωφορεία. Οχήματα 60 θέσεων που κυκλοφορούν τελικά με δύο-τρεις ανθρώπους, δύο-τρεις επιβάτες. Γίνεται λοιπόν ε, δημόσια ανάθεση και βλέπετε δεν έχει κανένα νόημα ε, να έχουμε τέτοια τεράστια οχήματα που ε, κυκλοφορούν με δύο-τρεις επιβάτες. Καλύτερα να υπήρχαν δύο-τρία αυτοκίνητα δηλαδή, να χρησιμοποιούσε ο καθένας το δικό του και δεν χρειάζεται συνεχώ να επιβάλλουμε νέα τέλη. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι αντιπαραγωγικό. Πρέπει λοιπόν να βελτιστοποιήσουμε τι μεταφορέ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Λούγκρεν. Εγώ έχω ζητήσει το λόγο και θα δώσω και ένα λεπτό στον κύριο Κράμερ στη συνέχεια. Γιατί κάνουμε αυτή τη συζήτηση σήμερα για την Ευρωβινιέτα, το Ευρωπαϊκό Τέλος Κυκλοφορίας. Αυτό είναι το βασικό ζήτημα. Επειδή ο κόσμος αλλάζει. και αλλάζει ο κόσμος επειδή έχουμε τη ρήπανση που είναι η ασθένεια του 21ου αιώνα. Εφόσον θα έχουμε εκατοντάδε. χιλιάδες πρόωρους θανάτους στην Ευρώπη, τι θα κάνουμε. Βλέπουμε τα βαρέα οχήματα στα οδικά δίκτυα, οχήματα και υπερθυμίζω ότι στην πλειονότητα αυτών των οχημάτων υπάρχει μόνο οδηγός. Και δεν συμφωνώ, κ. Λούγκεν, που είπατε ότι χρειαζόμαστε βαρέα οχήματα, μεγάλα φορτηγά στους δρόμους. Εμείς λέμε ότι αυτά τα μεγάλα οχήματα, τα μεγάλα φορτηγά μπορούν να μπουν στο σιδηρόδρομο. Και αυτό θα μας επιτρέψει να καταπολεμήσουμε τη ρήπανση. Πρέπει λοιπόν να βοηθήσουμε τις χώρες να κάνουν αυτό και να αλλάξουν νοοτροπία. Και αυτή η αλλαγή νοοτροπίας είναι σημαντική. Δεν το λέω για μας αυτό. Εργαζόμαστε αυτή τη στιγμή και για τις επόμενες γενιές. Γιατί Ακόμα και όταν έχουμε εξάρσεις ρήπανση, τι θα λέμε δηλαδή, να μείνουν ηλικιωμένοι ε, στα σπίτια τους, τα παιδιά να μην πηγαίνουν στο πάρκο επειδή υπάρχει κίνδυνος για την υγεία τους, στις εγγύους να λέμε μείνετε σπίτι, τι κόσμος είναι αυτός. Επομένως, η οικολογική φορολογία θα πρέπει να αποτελέσει μια ευκαιρία για να αλλάξουμε τη ζωή μας. Ορισμένες φορές πράγματι αυτό είναι δύσκολο. Το πραγματικό ζήτημα λοιπόν είναι ότι θα πρέπει να εφαρμόσουμε την αρχή ορυπαίνων πληρώνει και θα πρέπει αυτή η αρχή να εφαρμόζεται παντού γιατί έχουμε και δεσμεύσεις ως προς το κλίμα. Το δεύτερο, τι είδους συλλογική ευφυΐα θα επιδείξουμε σε αυτά τα έσοδα. Και είχαμε τους Ελβετούς συναδέλφους εδώ και μας είπαν δείτε πώς λειτουργεί το σύστημα, δείτε πόσο έχουμε επενδύσει στο σιδηρόδρομο και πόσε θέσεις απασχόλησης ε, δημιουργούνται. Αυτοί δεν κάθονται τώρα να μίζερα να λένε να μας κοστίσει 2%-5%. Όχι, λένε ένα συγκεκριμένο ποσοστό πάει στις αναλυτικές μεθο... Ε, στους τρόπους μεταφοράς. Και βλέπουμε ότι αυτό λειτουργεί και από οικονομικής άποψης, αύξηση της απασχόλησης, αλλά και από πλευρά ανταγωνιστικότητα. Οπότε βγαίνουν όλοι κερδισμένοι. Έτσι πρέπει να δούμε τα πράγματα. Και κλείνω με το εξή. Η Ευρωβινιέτα δεν θα πρέπει να αποτελέσει περιορισμό για μας, αλλά ευκαιρία για να δείξουμε ότι η φορολογία δεν είναι μόνο για να τιμωρήσουμε τους ε, ρηπαίνοντες, απλώς ε, ως ευκαιρία θέλουμε να καταστήσουμε την ε, κινητικότητά μας κινητικότητα του 21ου αιώνα. Κύριος Κράμερ. Monsieur Wim van de Kamp, c'est Monsieur Kramer et après ça vous. Point of order. Comment Vous voulez me faire attaquer au tac. Allez-y. Als meneer Kramer een kort... Επίση διαδικασία. Αν ο κύριος Κράμερ έχει σύντομο ερώτημα, συμφωνώ να πάρει τον λόγο. Αλλά αν θέλει να δευτερολογήσει, τότε πραγματικά ενίσταμα. Ήθελα μόνο να το πω. Alors, Monsieur Kramer, votre question. Ερώτηση, κύριε Κράμερ. Δεν ήθελα να θέσω ερώτηση, ήθελα να επανέλθω. Γιατί απαγορεύεται να δευτερολογήσω, λέει ο κύριος Κράμερ. Ας συνεχίσουμε, ας συνεχίσουμε, μην χάνουμε χρόνο. Κύριε Κράμερ, ένα λεπτό με τις περιοχές της Υπέθρου. Εκεί τα νίκια είναι πολύ χαμηλά. Κανείς δεν συζητεί γι' αυτό. Όταν μπαίνει όμως διόδιο, το διόδιο δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε αύξηση. Και δεύτερο, στις 24 Βιμ, όταν θα έχουμε την ημερομηνία, αν παντρευτούμε και οι δύο, τότε ίσως ο Πέτερ Βαντάλεν να καταλήξει να έχει την πλειοψηφία. Να είναι καθαρό αυτό, ε. Σας ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα ας απαντήσει στις διάφορες παρατηρήσεις που έγιναν. Η κυρία Βέρνερ. Γενική Διεύθυνση ΜΟΥΒ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους και όλους. Είναι θαυμάσια η έκθεση και η κατεύθυνση που λαμβάνει η συζήτηση. Η, η συγκήτριά σας έδωσε σαφή υποστήριξη στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την πάει παραπέρα και ενισχύει τις βασικές αρχές της. Ε, χαιρόμαστε πολύ που βλέπουμε και το μεγάλο ενδιαφέρον που επιδεικνύει και η Επιτροπή Μεταφορών και Περιβάλλοντος αλλά και ε, η προστασία των καταναλωτών και για το φορολογικό μέρος του προτάσεώς μας. Για την επιβάρυνση, για το charging, η συγκίτρια προβλέπει να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής και σε μοτοσυκλέτες και στο δευτερεύον οδικό δίκτυο. Και αυτό για μας είναι θετικό, διότι θα οδηγήσει σε συνεκτική επιβάρυνση σε ευραίο πεδίο και επιτρέπει και στις χώρες μέλη να το κάνουν όταν θα θεωρήσουν ότι είναι εύθετος ο χρόνος και λόγω των συνθήκων που ισχύουν στις χώρες τους. Και για την μη διακριτική εφαρμογή σε διάφορες κατηγορίες οχημάτων και ιδίω η η εφαρμογή σε ελαφρά και μέσου βάρους φορτηγά αυτοκίνητα πρέπει να γίνει το δυνατόν συντομότερο. Χαιρόμαστε και με την ιδέα για την απαλλαγή των αυτοκινήτων οχημάτων που έχουν μηδενικές εκπομπές καυσαερίων. Τώρα, για τη χρήση των βινιετών γνωρίζουμε ότι είναι διαφορετικές οι προσδοκίες των χωρών μελών σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των συστημάτων. Ταυτόχρονα θα πρέπει να αναμένουμε από τις χώρες μέλη να ζητήσουν κάποια ευκαμψία στην εφαρμογή. Άρα θα πρέπει να συζητήσουμε ρεαλιστικές προθεσμίες. Κάποιες ομάδες προτείνουν επίσης τη δυνατότητα να περιληφθούν και εξωτερικό κόστος και ε, χρέος ή μάλλον ε, χρέωση ε, για τις συμφορήσεις, για τις εχμές κυκλοφορίας γίνει αλλαγές οι οποίες θα μας επιτρέψουν να προσεγγίσουμε στην εφαρμογή της αρχής ορυπαίνων πληρώνει, άρα καταρχήν είναι σωστή κατεύθυνση, αλλά θα πρέπει να δούμε ρεαλιστικά ποια από αυτά τα πράγματα είναι δυνατόν να δεχθεί και το Συμβούλιο Υπουργών. Όπως γνωρίζετε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υπέρ της επανεπένδυσης των εσόδων στον τομέα των μεταφορών. Μπορεί να πάνε δηλαδή σε πολυτροπικές μεταφορές στους σιδηροδρόμους, στην εγγύηση της ασφάλειας, αλλά και στη συντήρηση υφισταμένων ε, οδών. Πάντως η πρότασή μας ε, βλέπω ότι ιστερεί και απέναντι στις φιλόδοξες τοποθετήσεις των μελών της Επιτροπής σας. Χαίρομαι που βλέπω ευρεία υποστήριξη για τα μέτρα που αποσκοπούν στην καλύτερη αποδοχή από πλευρά του κοινού, δηλαδή αύξηση τη διαφάνεια για το πώ θα χρησιμοποιηθούν τα έσοδα από την φορολόγηση αυτή, από την επιβολή των διοδίων δηλαδή. Και τέλο, για, τα, για του ασφαλεί χώρου σταθμεύσεων στι ε, οδού που θα ε, έχουν διόδια, θα βοηθήσει και για την αποδοχή των διοδίων, αλλά και για την βελτίωση τη ασφάλεια των ε, οδών αυτών, καθώ και τη ασφάλεια των ίδιων των οδηγών υπάρχουν πολλές διασυνδέσεις που μπορούν να γίνουν μεταξύ των θεμάτων αυτών και θα δούμε και πώς θα συνδυάσουμε τις προτάσεις που συζητούμε σήμερα. Λίγα λόγια τώρα σχετικά με κάποιες από τις τροπολογίες που έχουμε δει και για να σας καταστήσω προσεκτικούς πρώτα για την ε, ουσιώδη αλλαγή σε καθεστώς διοδίων. Εμείς προτείναμε το πολύ 5% στην αλλαγή των εσόδων σε σύγκριση με τον προηγούμενο χρόνο εκτός πληθωρισμού. 5% είναι ήδη σημαντικό ποσό για τους χρήστες και πολλοί εξημών ζητήσατε μεγαλύτερη ευελιξία και αύξηση της ενδεχόμενης αυτής αλλαγής. Εμείς θεωρούμε ότι το 15% που προτείνει η συγκήτρια είναι μάλλον και το μέγιστο όριο που θα μπορούσε να προσεγγίσει κανείς και είναι ήδη υψηλότερο του 10% αλλαγής που περιλαμβάνεται στις, ε, στην οδηγία περί παραχωρήσεων. Και τέλος, η εφαρμογή τελείως διαφορετικών κανόνων στα, στα διόδια παραχωρήσεων είναι κόκκινη γραμμή για μας. Δεν θα πρέπει δηλαδή να δίνει αυτό το ελεύθερο στους παραχωρησιούχους να κάνουν ό,τι θέλουν. Όπως έχω πει και παλαιότερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει τη δυνατότητα να εφαρμόζονται κάποια ανώτατα ωραία, markup, αλλά θα πρέπει να δούμε ποια είναι ουσιώδης αλλαγή σε ρύθμιση επιβολής διοδίων. Χρειάζεται να υπάρχουν εύκαμπτοι κανόνες, αλλά τα markup σημαίνουν πάλι σημαντική αύξηση των διοδίων. Και οι χρήστες αναμένουν βέβαια και θεμητό είναι τα βάρη να είναι πάρα πολύ προσεκτικά υπολογισμένα. Επίσης, συμφωνούμε με το στόχο της προώθησης της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής και νομίζω ότι συνεχίζεται ένας καλός προβληματισμός που λέει μείωση ίσως κατά 50% υπέρ των ανθρώπων που κινούνται πάντα στην ίδια διαδρομή πηγαίνοντας από τη δουλειά στο σπίτι και ανάποδα. Και σε ό,τι αφορά τα αστικά κέντρα, το να μπει αυτό νομίζω ότι μπορεί να οδηγήσει στο αντίθετο αποτέλεσμα και να επιβαρύνει τις συμφορήσεις. Αν υπάρχει τρόπος να ελαφρυνθεί το βάρο για τους κομιούτερ, αυτό δεν θα πρέπει να ισχύει μόνο για τα αστικά κέντρα, αλλά και για απομακρυσμένε περιοχές όπου δεν υπάρχει εναλλακτική δυνατότητα μεταφοράς από την οδική. Τέλος, για, τα εξωτερικά, για το εξωτερικό κόστος των ατυχημάτων. Για μας δεν είναι σωστό να περιληφθούν τα έσοδα από τα διόδια. Καλύτερα να γίνει μέσω ασφαλίσεων ή φορολογικών επιβαρύνσεων οι αυτοκινητόδρομοι που έχουν διόδια είναι από τους πλέον ασφαλείς. Να καθίσουν το να πληρώνουν όλοι αυτοί για τα ατυχήματα στο συγκεκριμένο δρόμο νομίζω ότι δεν δικαιολογείται. Βεβαίως είμαστε διατεθειμένες να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα σε λεπτομέρεια. Και σας ευχαριστώ πάντως για τον γενικό προσανατολισμό της εκθέσεώς σας. Ευχαριστώ κυρία Βέρνερ. Θα δώσω το λόγο πάλι στην εισηγήτριά μας για να μπορέσει να τοποθετηθεί για τις διάφορες παρεμβάσεις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους σκιώδεις συζητητές και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς και τους άλλους ευρωβουλευτές που τοποθετήθηκαν. Έχετε δίκιο και απευθύνομαι εδώ ιδίω στον Ζορζ Ντομινίκ και την κυρία Γιούτο, δεν μίλησα για το earmarking και για την χρήση των εσόδων. Ίσως θα έπρεπε να είχαμε μιλήσει από την πρώτη συνάντηση των σχεδόν εισηγητών. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα. Και βέβαια νομίζω ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ευρεία συνένεση για το θέμα αυτό, που είναι πράγματι πολύ σημαντικό, για να ε, γίνει αποδεκτή το, αποδεκτό το σύστημα αυτό. Δεν τα είπα, εσείς καλά το είπατε, Συνεχίζω πάντως στην επόμενη συνάντηση των σχεδόν εισηγητών θα συζητήσουμε και το θέμα αυτό που είναι πράγματι απαραίτητο να γίνει αυτό. Σε ό,τι αφορά τις συμβάσεις παραχωρήσεων που επανήλθαν πολλές φορές. Ο τρόπος με τον οποίο θα εξήγησε ο Ντιμινίκ Κρικέ είναι σωστός. Δεν λαμβάνεται υπόψη σήμερα στις παραχωρήσεις αυτές η αρχή του Ολυπαίνων πληρώνει επ' αυτού του μέρους των συμβάσεων θα πρέπει να επέλθουν τροποποιήσεις. Είναι γνωστοί οι κανόνες παρόλα αυτά. Οι δύο αυτές αρχές που περιλαμβάνονται στο σχέδιο οδηγίας που δεν μπορούμε πλέον να την αποκαλούμε ευρωβινιέτ αλλά ευρωέσοδο ε, θα πρέπει να εφαρμόζονται. Για την ημερομηνία της ψηφοφορίας Συμφωνώ με την Πρόεδρο. Πρέπει να ψηφίσουμε οπωσδήποτε στις 24 Πέμπτου. Θυμίζω ότι εδώ και ένα χρόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε το πρώτο σχέδιο για το πακέτο της κινητικότητας, το οποίο αναμέναμε με ανυπομονησία για να μπορέσουμε να εργαστούμε. Και νομίζω ότι το σύνολο των σχεδόν εισηγητών είναι διατεθειμένες και διατεθειμένοι να εργαστούν όσο χρειάζεται για να καταλήξουμε σε ένα στέρεο κείμενο που να μπορέσει να ψηφιστεί στις 24 Πέμπτου. Και βεβαίω στι συνεδριάσει των επιτροπών είναι και παρόντε οι ευρωβουλευτέ, άρα δεν με ανησυχεί. Ένα θέμα το οποίο έφυξαν διάφοροι συναδελφοί μου για το δευτερεύον οδικό δίκτυο που προτείνεται να περιληφθεί στο πεδίο εφαρμογή αυτό να μην έρθει από πάνω και να περιλάβει όλο, όλο το δευτερεύον οδικό δίκτυο. Θα πρέπει χώρες μέλη ή οι τοπικές αρχές να αποφασίσουν αυτές που είναι αρμόδιες για να μπορέσουν να επεκταθούν. Δηλαδή δεν είναι ανάγκη να είναι από το ένα χωριό στο άλλο. Αλλά το δευτερεύον οδικό δίκτυο που γνωρίζουμε ότι στην πραγματικότητα τμήματά του χρησιμοποιούνται για να αποφεύγεται η κυκλοφορία πάνω σε αυτοκινητοδρόμους που επιβαρύνονται με διόδια. Οι δύο αρχές Χρήστη πληρώνει, ρηπαίνων πληρώνει, ναι μεν ναι, θα εφαρμόζονται, αλλά δεν σημαίνει ότι όλοι οι ευρωπαϊκοί δρόμοι θα αφορώνται από την συγκεκριμένη ρύθμιση. Καθόλου δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο και θα πρέπει να είναι βέβαιο. Για όσον αφορά την συμπερίληψη των δημοσίων μεταφορών, δηλαδή λεωφορεία και πούλμαν, τα συζητήσαμε πολύ στην πρώτη συνάντηση των σχεδόν εισηγητών. Θα πρέπει να βρεθούν κάποιε ρυθμίσει, Πάλι όμω δεν υπάρχουν εξαιρέσεις. Από την αρχή χρήστης πληρώνει, ρηπαίνων πληρώνει. Λαμβάνεται όμως υπόψη η χρήση της οδού που γίνεται και ιδίω για τα λεωφορεία που επιτρέπουν να μετακινηθεί ο επιβάτης στο τελευταίο εκείνο ε, διάστημα, στη τελευταία εκείνη απόσταση που δεν καλύπτεται ας πούμε από τον σιδηρόδρομο. Θα πρέπει να σεβαστούμε το χρονοδιάγραμμα, να έχουμε μια στέρεα συμφωνία μεταξύ μας και ευχαριστώ όλες και όλους τους κοιόδης για τη συνεργασία τους. Σας ευχαριστώ κυρία Συγγήτρια για το κείμενο λοιπόν, για το ευρωέσοδο. Θα η ευρωτέλος 24 Πέμπτου στις 9 το πρωί η ψηφοφορία για το κείμενο. Να συνεχίσουμε τώρα για την φορολογία οχημάτων. Θα λάβει το λόγο η κυρία Κλούνε και μετά οι υπόλοιποι συνάδελφοι που επιθυμούν να λάβουν το λόγο και μετά θα παρακαλέσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κυρία Κλούν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως είπαμε, αυτός ο φάκελος σχετίζεται άμεσα με το θέμα που μόλις συζητούσαμε, επιβολή των τελών και ο τρόπος της επιβολής, ανάλογα με την χρήση των δρόμων, φορολόγηση, υψηλή φορολόγηση. Συνδέονται λοιπόν άμεσα αυτά τα θέματα και με την πρόταση της Κομισιόν για την ε, διευκόλυνση των χώρων μελών. ώστε να δούμε υπόψη μας και τα HGVs, τα οχήματα αυτά, τα βαρέα. Προτείνεται μια πενταετία ως περίοδος εφαρμογής. Θα ήθελα να υπάρχει όμως απλούστευση και να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία ώστε να λάβουμε υπόψη μας το διοικητικό βάρος για τις χώρες μέλη και να λάβουμε υπόψη μας και τις διαφορετικές εθνικές ιδιαιτερότητες όσον αφορά το τέλος και την επιβολή του σε σχέση με αυτά που προτείνει η Κομισιόν. Να πω καταρχάς επίσης ότι είμαι σύμφωνη με την αρχή της επιβολής του τέλους ανάλογα με την απόσταση και όχι το χρόνο. Είναι σημαντικό το θέμα λοιπόν να το έχουμε κατά νου για διάφορες χώρες μέλη Οπότε οι χώρες μέλη πρέπει να έχουν την ευελιξία να μειώσουν ή να απαλείψουν τέλη αν ε, θεωρούν ότι είναι απαραίτητο. Οπότε θα πρέπει να υπάρχει αυτή η δυνατότητα να τους δίνουμε λοιπόν περισσότερη ευελιξία. Είχαμε 41 λοιπόν τροπολογίες που καλύπτουν διάφορα ζητήματα και κάποιες από αυτές τονίζουν και υπογραμμίζουν την ανάγκη το να δοθεί ευελιξία στην επιβολή στις χώρες μέλη. Επίσης ε, για τον άνθρακα θα πρέπει να το συζητήσουμε κατά πόσο αυτό εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογή. Θα το δούμε σε μια συνάντηση των σκιωδών. Συνολικά όμως από τις τροπολογίες βλέπουμε ότι είναι σημαντικό να υπάρχει, ξαναλέω, δυνατότητα ευελιξία στις χώρες μέλη. και επιβολή τελών, ιδιαίτερα για τα βαρέα οχήματα και κατά πόσο αυτή βέβαια θα έχει επιπτώσει στι μικρομεσαίε επιχειρήσει σε σχέση με το θέμα που συζητούσαν προηγουμένω για την χρήση των δρόμων. Για τι μικρομεσαίε θα πρέπει να δούμε την δομή των δρόμων και τη υποδομή στην Ευρώπη. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν κατά πόσο χρησιμοποιούνται συγκεκριμένοι δρόμοι από βαρέα οχήματα για τη μεταφορά αγαθών, γιατί αυτό είναι σημαντικό. Αυτά από μένα. το συνδέουμε με το προηγούμενο ζήτημα αυτό και θα είμαστε έτοιμοι νομίζω να, να ψηφίσουμε στις 21 του Μάη και ξαναλέω από το βλέμμα των τροπολογιών συμφωνούμε και με τη δική και με αυτή της Κομισιόν και φαντάζομαι ότι θα έχουμε μια συμφωνία, μια να ψηφίσουμε και για το επόμενο σημείο στις 24 του Μάη. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Κλούν, λέει Πρόεδρο, Όχι 21 όμω 24 έτσι, όχι 21, 24. Θα το ξαναπώ δύο-τρεις σήμερα για να το εμπεδώσετε. 24. Ναι, εγώ είπα πρόεδρε 24 όμως. Γιατί 21 άκουσα εγώ. 24, 24, έτσι. Κάντε ό,τι θέλετε, κάντε ό,τι θέλετε, αλλά 24 να είστε ελεύθεροι 9 ε, η ώρα εδώ. Ξεκινάμε τη συζήτηση λοιπόν. Ευχαριστώ κύριε Κλούν για τι ε, θέσει σα. Κύριε Ταπαρντέλ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Να πω και εγώ ότι ευχαριστώ την εισηγήτρια και ω ε, σκιώδη εισηγήτρια των εισηγητών. Θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πράγματι χρειάζεται ένα σύστημα μεταφορών αποτελεσματικό, αξιόπιστο, που θα ανταποκρίνεται στις περιβαλλοντικές και άλλες προκλήσεις. Ναι, εδώ μιλάμε πραγματικά για την επιβολή τελών ως ένα στοιχείο ανάλογα με την απόσταση και μιλάμε για την ετήσια επιβολή τελών. Και είναι αλήθεια ότι οι στατιστικές μας δείχνουν σήμερα ότι αυτά τα τέλη δεν αντανακλούν την πραγματική χρήση των υποδομών και δεν είναι αποτελεσματικά τα τελευταία σαν αφορά τη μείωση των ρήπων. Οπότε θα πρέπει μέσω μακροπρόθεσμα να έχουμε στόχο τη μείωση των τελών που ήδη επιβάλλονται σε διάφορες χώρες μέλη. Και μάλιστα τη στιγμή που οι επενδύσεις αυξάνονται στις υποδομές. Πάντω να ευχαριστήσω, μάλλον να επιστήσω την προσοχή τη Κομισιόν και της ε, εισηγήτρια σε κάποιου κινδύνου. Δηλαδή έχουμε κάποια μέτρα τα οποία πραγματικά προωθούν κάποιε μορφέ μεταφορών μειώντα το συνολικό κόστο, όμω η μείωση τελών αναόχημα θα μπορούσε να έχει αρνητικέ επιπτώσει όσον αφορά του προπολογισμού των τοπικών, περιφερειακών και εθνικών αρχών. Οπότε θα πρέπει συγκεκριμένα εδώ να δούμε πριν κάνουμε αλλαγέ στην ε, φορολογία να έχουμε μια βαθμιαία προσέγγιση ώστε να υπάρχει ευελιξία και για να θεσπίσουμε βέβαια και ταυτόχρονα και την απαραίτητη αυτή αρχή, δηλαδή τη επιβολή τελών ανά απόσταση. Και από ό,τι βλέπω, αυτή είναι και η γενική προσέγγιση όλων των εισηγητών σε αυτό το φάκελο. Πάντω είμαστε έτοιμοι, θα είμαστε έτοιμοι στι 24 του Μάη για να υιοθετήσουμε την έκθεση αυτή. Ευχαριστώ. Κύριε Ερικέ, έχετε το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομος. Καταρχάς να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τα δουλειά της και υπάρχει γνήσια και πραγματική ευθυγράμμιση μεταξύ της πρότασης της Κομισιόν, της στάσης της εισηγήτριας και της πλειοψηφία των ε, σκιωδών και συνεισηγητών. Εμείς θα θέλαμε βεβαίως να υπάρχει και συνάφεια και με την προηγούμενη οδηγία δηλαδή την ε, οδηγία για αυτά τα έσοδα που αφορούν τις μεταφορές. Η συνάφεια λοιπόν είναι λέξη κλειδί εδώ και μετά. Μετά από αυτά που είπε η συγγήτρια θα έπρεπε να κάνουμε πιο ομοιογενείς τις διαφορές φάσεις. γιατί όντως ε, υπάρχει ο κίνδυνος καθυστέρησης και περιπλοκότητας για την ε, κάθε αλλά και για τους χρήστες. Οπότε θα πρέπει όλα αυτά να γίνουν πιο ομοιογενή. Και θα πρέπει επίσης η τεχνική εναρμόνιση να είναι ευανάγνωστη μεταξύ των διαφόρων διατάξεων. Η πρόταση λοιπόν της Κομισιόν είναι ενδιαφέρουσα έκθεση αυτή νομίζω τελικά δεν έχει δεχτεί πάρα πολλέ τροπολογίες, οπότε θα πρέπει να είμαστε ευθυγραμμισμένοι με αυτά που κάνουμε για αυτά τα έσοδα που λέγαμε προηγουμένως και θα πρέπει να θεωρούμε βέβαια την αρχή ο πληρώνει. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας βέβαια και τις οικονομικές ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά θα πρέπει να είμαστε ε, συνεπείς επίσης και με αυτό το πλαίσιο το φορολογικό που αφορά το περιβάλλον. Αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ρικέ. κύριο Κράμερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομοθετική, ε, μάλλον φορολογική νομοθεσία δεν είναι αρμοδιότητα της Ένωσης αλλά των χωρών μελών. Και γνωρίζουμε βέβαια ότι οι χώρες κάνουν και πολλές ανοησίες στην φορολογική νομοθεσία. Ε, είμαι Γερμανός, όλοι έχετε ακούσει για το σκάνδαλο του Ντίζελ. Όμως, ενώ γνωρίζουμε για την μεγάλη ε, ζημιά που κάνουν λόγω ρήπανσης 600.000 πρόωροι θάνατοι στη Γερμανία λόγω των ε, οξυδιών του αζότου. Και όμως, και όμως επιχορηγείται από τον δημόσιο προϋπολογισμό το καύσιμο ντίζελ. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την παρουσίαση του θέματος καθώς και για τη συνεργασία μαζί μας. Εμείς θα κάνουμε μια πρόταση. Εάν πρόκειται να επιβληθεί η φορολογική επιβάρυνση θα πρέπει να ληφθούν υπόψη διάφοροι παράγοντες μεταξύ αυτών και το βάρος του οχήματος. Σας είπα για το ντίζελ ο κινητήρας δίζελ χρειάζεται κάπως λιγότερα καύσιμα από τη βενζίνη. Γι' αυτό και άρχισε πριν από 30 χρόνια η επιδότηση του καυσίμου δίζελ. Επειδή όμως ήταν τόσο υψηλή η επιδότηση, τα αυτοκίνητα αυτά έγιναν όλο και βαρύτερα και μεγαλύτερα. Και τελικώς ο απολογισμός βγαίνει αρνητικός, ενώ αρχικά ήταν θετικός. Γι' αυτό λέμε να ληφθεί υπόψη το βάρος στη φορολόγηση των αυτοκινήτων και βέβαια οι εκπομπές διοξιδίων ε, του ανθράκου, αλλά και οι εκπομπές σωματιδίων ε, και οξυδίων του αζότου. Λίγο παραπάνω χρήματα για να αποκτήσει κανείς ένα πιο καθαρό αυτοκίνητο και να προστατεύσει έτσι το περιβάλλον και ιδίως την υγεία των συνανθρώπων δεν θα πρέπει να ε, επιβαρύνεται. Όποιος όμως θέλει ντε και καλά ένα μεγάλο πολυτελές και ρηπογόνο αυτοκίνητο ε, να, επιβα... να επιβαρύνεται λίγο περισσότερο. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι κάπως δύσκολο να ε, συναρμοστούν όλα αυτά, αλλά καλό θα είναι στη συζήτηση να διαρευνηθούν όλες οι δυνατότητες. Σε ευχαριστώ κύριε Κράμερ. Κύριε Λούντγκρεν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ενδιαφέρον. Γιατί θυμάμαι ότι ήδη είχαμε συζητήσει ότι θα πρέπει να προσέχουμε το περιβάλλον, θα πρέπει να είμαστε οικολόγοι, θα πρέπει να παράγουμε περιβολικό διοξείδιο του άνθρακα κλπ. Εγώ ομολογώ ότι θέλω να προστατεύσω το περιβάλλον, αλλά μου αρέσουν και οι βόλτες με το αυτοκίνητο. Και εκεί που μένω εγώ, μόνη μετακίνηση που είναι δυνατή είναι με το αυτοκίνητο. Ίσως θα πρέπει να θυμάμαστε ότι υπάρχουν πάρα πολλά αυτοκίνητα τα οποία δεν ρηπαίνουν και τόσο. Οπότε ενδεχομένω θα έπρεπε να αρχίσουμε να εμπνεώμαστε με τα παραδείγματα αυτών των ανθρώπων πραγματικά που οδηγούν αλλά χωρίς να ρηπαίνουν. Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας ανταγωνισμός μεταξύ των διαφόρων μορφών μεταφορών. Δυστυχώς όμως λείπουν οι αποδείξεις καμιά φορά. Σε σχέση δηλαδή με το να έχουμε ας πούμε πιο ασφαλείς και πιο ταχύς σιδηροδρόμους ας πούμε. Στη Σουηδία Εμεί έχουμε τεράστιε εκτάσει δασικέ. Εκεί λοιπόν δεν μπορούμε να επιβάλλουμε στον κόσμο πώ να μετακινείται. Δεν μπορούμε δηλαδή υποχρεωτικά να ας πούμε χρησιμοποιήσετε τον σιδηρόδρομο γιατί δεν γίνεται σε αυτές τις περιοχές επειδή δεν υπάρχει εναλλακτική λύση στο αυτοκίνητο. Οπότε εντάξει, σωστό να λέμε ότι ε, θα πρέπει να χρησιμοποιούμε τα δημόσια μέσα, το σύνδρομο κτλ. Αλλά αν υπάρχουν αναλλακτικέ, αν δεν υπάρχουν, τι να κάνουμε και στις μεταφορές εμπορευμάτων επίσης. Βεβαίως θα χρησιμοποιήσουμε το σιδηρόδρομο και άλλα. Αλλά όπου γίνεται. Και πρέπει να λάβουμε υπόψη μας επίσης και την σωστή συντήρηση των υποδομών. Δηλαδή, οι υποδομές να σε καλή κατάσταση για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν. βλέπω ότι αυτά που λαμβάνουμε α, ως έσοδα από τα τέλη καλύπτουν τρύπες του προπολογισμού. Και τώρα να στραφώ προς την Κομισιόν. Κομισιόν, ναι, ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι πολύ σύντομη. Πολύ σαφής η έκθεση και οι τροπολογίες Ξέρετε βεβαίω ότι η φορολόγηση είναι ένα θέμα ευαίσθητο για τις χώρες μέλη, αλλά συμφωνούμε ότι θα πρέπει βεβαίως να τηρηθούν οι στόχοι της Κομισιόν και να υπάρχουν μειώσεις με ένα βήμα, με μια πράξη. Πολύ ωραία, αλλά βέβαια εντάξει, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα για τις χώρες μέλη να το κάνουν αυτό νωρίτερα από πριν δηλαδή από το 24, ίσως από την ε, εφαρμογή της οδηγίας. Αυτό είχα να πω μόνο. Βεβαίως όλα αυτά σχετίζονται άμεσα με την, με την έκθεση που συζητήσαμε προηγουμένω. Να έχουμε λοιπόν πάντοτε παρόντες στο μυαλό μας τους ο, στόχους και να δούμε ακριβώ θα γίνει στη συνέχεια στο Συμβούλιο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Βέρνερ. Κυρία Κλούν, εσείς κλείστε το. Ευχαριστώ. Να υπάρχει συνένεση και καλή διάθεση. Να πω πάντως ότι η φορολόγηση είναι ένα θέμα σημαντικό για τις χωρίς μέλη. Οπότε, αν το και έχουμε την διαβούλευση, θα πρέπει το Συμβούλιο να λάβει υπόψη την άποψη του Κοινοβουλίου. Είτε δεσμεύεται είτε όχι από αυτήν. Εμείς λοιπόν γνωμοδοτούμε εδώ και το Συμβούλιο θα πρέπει να το λάβει υπόψη του. Πάντως, νομίζω ότι υπάρχει προσέγγιση και θα έχουμε νομίζω πολύ καρποφόρες συναντήσεις με τους σκιώδες τους επόμενους μήνες. Πάντως ευχαριστώ και τους σκιώδες αλλά και την Κομισιόν της Συμβουλή σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Κλούν, υπενθυμίζω ότι η ψηφορία θα στις 24-24 του Μάη 9 η ώρα το πρωί. Κύριε Σαλίνη, καλημέρα. Περνάμε σε εσά. Διαλειτουργικότητα των συστημάτων τηλεδιοδίων κλπ. Σας δίνω το λόγο και μετά θα ακούσουμε και τους σκιώδεις και όσους θέλουν να συμμετάσχουν στη συζήτηση. Παρακαλώ κύριε Σαλήνη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Η λόγω έκθεση αναφέρεται στη σωστή απόφαση εκ μέρους της Κομισιόν για αναθεώρηση μιας οδηγίας, δηλαδή αυτής για τα τηλεδιόδια, που παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα εφαρμογής. Οπότε η Κομισιόν προτείνει δύο στόχους που εμείς βεβαίω συμμεριζόμαστε, τουλάχιστον εγώ προσωπικά. Για την εσωτερική μας συζήτηση Κοινοβούλιο αφενός ένα στόχο είναι η προσπάθεια να εναρμονίσουμε επιτέλους τα συστήματα τηλεδιοδίων πανευρωπαϊκά, δηλαδή την τεχνολογική πτυχή. Ξέρουμε ότι υπάρχουν διάφορες τεχνολογίες στα πλαίσια αυτή τη παροχή υπηρεσία. Οπότε θα πρέπει να εντοπίσουμε ένα κριτήριο εναρμόνιση για τη χρήση, ώστε να υπάρχει διαλειτουργικότητα, η οποία όμως θα πρέπει να επιδιώκει και ένα δεύτερο βασικό στόχο, δηλαδή την ε, μείωση του αντικτύπου που παρουσιάζει σήμερα προβλήματα της μη πληρωμής από μια χώρα σε άλλη. Και στο μέτωπο αυτό, ιδιαίτερα για τη δικασία follow-up, για τις πληρωμές, έχουμε ακόμα και σήμερα ένα μεγάλο αριθμό νομικών προβλημάτων που σχετίζονται με την ε, δυνατότητα ενός εμπλεκόμενου, ενός φορέα στις μεταφορές στο αυτοκινητόδρομο σε περίπτωση που δεν πληρώνει τέλη σε άλλη χώρα ώστε να παραδίδονται τα στοιχεία του και να του ζητείται η καταβολή των τελών. Αυτή η έλλειψη λοιπόν η νομική Νομίζω αντισταθμίζεται από αυτή την παρήμβαση, την πολύ ικανοποιητική εκ μέρου τη Κομισιόν, συγκεκριμένα αναφέρουμε στα άρθρα 5 και 6. Υπάρχει λοιπόν και μία πτυχή που αφορά την τεχνολογία με ένα θετικό σημείο κίνηση. Παρ' όλα αυτά έχουμε διατυπώσει κάποιε παρατηρήσει κατευθείαν από το πρώτο προσχέδιο που πρότεινα και επέβαλα στους σκιώδεις εισηγητές και στις διάφορες τροπολογίες. Καταρχάς έχουμε το πολυτεχνικό ζήτημα που αφορά τις συχνότητες. Εμείς σήμερα έχουμε συστήματα και η Κομισιόν προτείνει σε σχέση με την πλατφόρμα των τηλεδιοδίων τις συχνότητες που σχετίζονται με τα ευφυή συστήματα μεταφορών και εδώ προτείνει η Κομισιόν μια μετάβαση από τα 5,8 GHz στα τηλεδιόδια στα 5,9 GHz που αφορούν ακριβώς αυτά τα ευφυή συστήματα μεταφορών. Εμείς συζητήσαμε τα θέμα εσωτερικά και με τους σκιώδες και υπάρχει μια διάχυτη αρνητική αξιολόγηση αυτής της ε, πρότασης επειδή τα κόστη απορρόφησης αυτής της μετάβασης θα είναι υψηλότερα από τα ωφέλη. Οπότε πρέπει να υπάρχουν περισσότερες δυνατότητες, περισσότερο ενδιαφέρον και ρεαλισμός για να προβλέψουμε την 5-8 συχνότητα, αλλά και ταυτόχρονα να αναζητήσουμε παράλληλα άλλες λύσεις τεχνολογικές με συστήματα που θα αποτρέπουν τις παρεμβάσεις, ε, παρεμβάσεις. Επίσης για το σήμα ER. Είχαμε διαφωνίες μεταξύ των σκιωδών και δεν απαραίτητο να συνεχιστεί αυτό θα βρούμε μια λύση. Πάντως η δική μου αρχική πρόταση ήταν να αξιολογήσουμε τις, την απόδοση της επιδόσης του MPR, του συστήματος συγγνώμη, MPR σε σχέση με τα τηλεδιώδια. Ο σύστημα εφαρμογής έχει ευρία χρήση σήμερα και είναι πάρα πολύ χρήσιμο το MPR για να στηρίξουμε άλλες τεχνολογίες τηλεδιοδίων. Όμως ω σύστημα άμεσης ε, συλλογή των ε, διοδίων παρουσιάζει με τη χρήση του σε διάφορες χώρες ένα επίπεδο αξιοπιστίας χαμηλότερο σε σχέση με τα υπόλοιπα τρία τεχνολογικά συστήματα που εξάλλου και η Κομισιόν έχει προβλέψει, έχει προτείνει. Οπότε θα πρέπει να κανονίσουμε εδώ αφενός αν υπάρχουν συνθήκες για να διασφαλίσουμε την ίδια αξιοπιστία Οπότε σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει το ενδεχόμενο να περιληφθεί στις υπόλοιπε τεχνολογίες. Διαφορετικά θα ήταν κάπως αντιφατικό αυτό, δηλαδή να εξισώσουμε αυτό το σύστημα, σύστημα ανάγνωσης δηλαδή ε, των πινακίδων με άλλα συστήματα, προηγμένα συστήματα, γιατί ε, ένας από τους στόχους ανθεώρησης της οδηγίας είναι ακριβώς το να μειώσουμε την μη καταβολή τελών. Οπότε είναι ξεκάθαρο θα πρέπει να ξεκινήσουμε από τεχνολογίες που ιδιαίτερα στο θέμα, στο θέμα των πληρωμών ήδη σήμερα παρουσιάζουν ψηλό επίπεδο και ψηλό βαθμό αξιοπιστίας. Τρίτο τεχνικό σημείο, τεχνικονομικό, αφορά την πρόταση περίληψης που υπέβαλε η Κομισιόν του καταλόγου τεχνολογιών σε ένα παράρτημα του διατακτικού και υπάρχει μια γενική αποδοχή με κάποιες διαφοροποιήσεις, αλλά υπάρχει τέλο πάντων πλειοψηφία των συναδέλφων σχεδόν εισηγητών που συμφωνούν μαζί μου ότι αυτός ο κατάλογος αποτελεί ένα ουσιώδες τμήμα της ε, οδηγίας και θα πρέπει να παραμείνει στο διατακτικό και όχι σε μια της πράξη. Παρ' όλα αυτά προτείναμε και καταθέσαμε στην τροπολογία 139 την δυνατότητα να εγκριθούν πιλωτικά προγράμματα τα οποία αφορούν τις νέες ε, τεχνολογίες που δεν θα προβλέπει η οδηγία. Ως χειρονομία αυτό, γιατί ξέρουμε ότι ο στόχος της παρέμβασης της Κομισιόν είναι το να προτείνουμε ένα ταχύτερο σύστημα σε σχέση με τον κατάλογο των τεχνολογιών, αλλά είμαστε πεπισμένοι ακόμα και στα πλαίσια της ε, συναπόφασης θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε τον πυρήνα τη οδηγία άθικτο και να τηρήσουμε ε, χρόνους παρέμβασης αποτελεσματικούς όσον αφορά τι υπόλοιπε τροποποιήσει. Ένα τελευταίο ζήτημα τεχνικού χαρακτήρα αφορά την δυνατότητα που ανέφεραν ε, κάποιοι συνάδελφοι να περιληφθεί δηλαδή στο διατακτικό και το θέμα των αστικών τελών, αστικών διοδίων. Η Κομισιόν κατά την άποψή μου δεν έχει περιλάβει για σωστούς λόγους τα τελευταία τα αστικά στην οδηγία γιατί νομίζω ότι ε, νομικά το υπόβαθρο των διοδίων στους αυτοκινητόδρομους, ε, στις σύραγγες κτλ. Ο προπολογισμό είναι τελείως διαφορετικός και οι προποθέσει που σε σχέση με τα αστικά τα τέλη. Και όπως είπαν διάφοροι συνάδελφοι στην συνάντηση των Σκιωδών, το να εξισώσουμε τα συστήματα αστικών τελών με το σύστημα τελών αυτοκινητοδρόμου θα προκαλούσε τεχνικά προβλήματα και κόστη που θα επιβαρύνουν τις τοπικές αρχές και αυτό δεν έχει υπολογιστεί ακόμα. Οπότε θα θέσουμε σε κίνδυνο που δεν έχει υπολογιστεί τις αρχές αυτές. Βέβαια έχουμε και τεχνικά προβλήματα και νομικά προβλήματα λοιπόν, τα οποία κατά την άποψή μου τίνουν στην διατήρηση αυτών των τελών, των αστικών, εκτός οδηγία. Αλλά βέβαια παραμένει ανοιχτή, ανοιχτό το ζήτημα προ συζήτηση. Υπάρχει ένα τελευταίο στοιχείο, το οποίο κατά την απόψή μου και στη συνάντηση των σχεδόν αναφέρθηκε και συζητήθηκε σημαντικά, ένα κύριο ζήτημα και είναι αντικείμενο πολλών τροπολογιών. Δηλαδή, η μεταφορά ενός σημαντικού τμήματος του περιεχομένου, περιεχομένου στο σημερινό προσχέδιο στο πεδίο των αποφάσεων της οδηγίας. Δηλαδή υπάρχουν διάφορα στοιχεία τα οποία δεν φαίνεται να είναι καθαρά τεχνικά αλλά είναι ουσιώδη και πρέπει να πω ότι υπήρξε θαυμάσια συνεργασία με την Κομισιόν επ' αυτού και μαζί αποτιμούμε πόσα και ποια στοιχεία αυτής της απόφασης θα πρέπει να προληφθούν στην οδηγία. Ε, για παράδειγμα, στο άρθρο 2, στους ορισμούς, όπου έχουμε νέους ορισμούς, παροχός, ε, ε, καταλότητα για χρήση κτλ. κτλ. Είναι πολλά αυτά. Μετά, πάντα για τα στοιχεία της απόφασης που θα πάνε στην οδηγία έχουμε όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις σε σχέση με τους ε, παρόχους αυτών των ε, υπηρεσιών, υποχρεώσεις τους, ε, εξαιρέσεις για τα διόδια κλπ. Και τέλος, επειδή για αυτό το ζήτημα υπάρχουν σημαντικά στοιχεία, κάτι το οποίο υποστήριξαν και τόνισαν και άλλοι συνάδελφοι σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων, αναμένουμε την νομοδότηση της ΛΥΜΠΕ, της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ, η οποία βεβαίως θα επικεντρωθεί στο θέμα της προστασίας των ευαίσθητων δεδομένων για να διαβάσουμε μετά, να κυκλοφορήσουμε τις συμβαστικές προτάσεις. Στις 19 του Απρίλη θα έχουμε την επόμενη συνάντηση των ε, ε, σχεδόν και για την εισήγηση αυτή, για την έκθεση με αυτή, προβλέπεται πάλι ψηφοφορία στις 24 του μήνα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Σαλήνη. Α περάσουμε τώρα στη συζήτηση. Η συνάδελφος Σενάλοβα έχει το λόγο πρώτη. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Πολύ σύντομα. Σε ό,τι αφορά τις παρατηρήσεις του εισηγητή, κατά τη διάρκεια της ε, συνάντησης των σχεδόν εισηγητών, νομίζω ότι η συζήτηση παίρνει πλέον μια καλή κατεύθυνση για τις λεπτομέρειες μπορώ να πω ότι συμφωνούμε σε πολλά σημεία. Για παράδειγμα, η συχνότητα να παραμείνει στα 5,8 GHz. Επίσης, συμφωνούμε ότι ο κατάλογος των τεχνολογιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τα ε, να συμπεριληφθεί στο διατακτικό. Ωστόσο, πρέπει να συζητήσουμε περαιτέρω σε ό,τι αφορά την οδηγία και τη δυνατότητα ε, ανάκτησης ε, των ε, διαφυγών των κερδών από τα τελεδιώδια. Ένα άλλο θέμα συζήτησης αφορά την αυτόματη ανάγνωση των πινακίδων κυκλοφορίας που θα μπορούσε να απλοποιήσει το σύστημα και των τηλεδιοδίων και της ανάκτησης των εσόδων. Νομίζω ότι η σε πολύ σωστά συνόψεσε τη συζήτηση. Δεν θέλω λοιπόν να επεκταθώ περαιτέρω. Ήθελα μόνο να σταθώ στα κέρια ζητήματα όπου ακόμα πρέπει να υπάρξει περαιτέρω εξέταση. Τον ευχαριστώ πάντως για το ανοιχτό του πνεύμα και θέλω να συνεχίσουμε αυτή την αγαστή συνεργασία. Ευχαριστούμε κύριο Στελίντσικα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Παίρνω το λόγο εξ ονόματο του συναδέλφου Βαν Μιλτέμπουργκ, που δυστυχώ ε, δεν μπορούσε να είναι εδώ σήμερα. Έχει συνάντηση με του κοιότητε συζητητέ ε, λόγω τη έκθεση που έχει αναλάβει στην ε, Επιτροπή Ρέτζι. Ήθελα λοιπόν να μεταφέρω ορισμένε από τι παρατηρήσει του. Κάποια βασικά στοιχεία που πρέπει να μεταφερθούν από, το, από την απόφαση της ETIS στην οδηγία ETIS για λόγους κοινής λογικής για να αποφύγουμε πιθανές αλληλεπικαλύψεις ε, στο κείμενο και ενδεχομένως ε, έλλειψη ασφαλές δικαίου. Ο κατάλογος των τεχνολογιών θα πρέπει να μπει στο παράρτημα και όχι στο διατακτικό του κειμένου. Η ευελιξία ε, απαιτείται για να προσαρμοστούμε στις τεχνολογικές εξελίξεις και να μην τις παρεμποδίζουμε. Φαντάζομαι συμφωνείτε προς αυτό είναι τεχνική απόφαση και όχι πολιτική απόφαση. Επομένω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να λάβει την εντολή να το διευθετήσει και η συμπερίληψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτή την περίπτωση οδηγεί μόνο σε ε, περιττό διοικητικό άκτο και καθυστερήσει. Η αυτόματη ανάγνωση των πινακίδων είναι καλό εργαλείο για τα τηλεδιόδια και διευκολύνει τη διασυνορική συνεργασία. Γι' αυτό εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογή τη ε, οδηγία αυτή, όπω προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτά θέλω να πει ο συνάδελφο για την πρόταση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Τελίνσκα. Το λόγο έχει ο κύριος Νταλούντε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Έχω τις εξή παρατηρήσεις. Πρώτον, χρειαζόμαστε ένα πλαίσιο το οποίο ε, να μην αφορά μόνο τα δικά δικτύα, αλλά και τις πόλεις μας. Γιατί ένα και προσθέτερες πόλεις εισάγουν τέτοια ε, συστήματα διοδίων. Και αυτό είναι πλέον κάτι το οποίο απασχολεί τους πολίτες που ε, ταξιδεύουν καθημερινά, πηγαίνουν στη δουλειά τους από τη μία πόλη στην άλλη, μπορεί από τη μία χώρα στην άλλη ενδεχομένω. Είναι λοιπόν σημαντική διαλειτουργικότητα. Μετά, οι πληροφορίες που συλλέγονται θα πρέπει να ε, χρησιμοποιούνται μόνο για το σκοπό για τον οποίο έχουν ε, συλλεχθεί. Και μετά, σε την αρχή, ο ρηπαίνων πληρώνει. Θα πρέπει τα διόδια αυτά να συμβάλλουν στην ολοκλήρωση ενός βιώσιμου συστήματος για, να έχουμε τελικά λιγότερη κίνηση στους δρόμους και λιγότερα σημεία συμφόρησης. Ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή για την πολύ καλή συνεργασία. Παρακαλώ, κύριε Λούνγκερ, θέλετε να πάρετε το λόγο. Όχι. Να δώσουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κυρία Βέρνερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Σαλίνη για την ευρεία στήριξη ε, προς την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι ιδιαίτερα τεχνική αλλά και εξίσου σημαντική για την ψηφιοποίηση και τη διαλειτουργικότητα των διοδίων. Το 1 τρίτο των τροπολογιών αφορά το βασικό ζήτημα της μεταφοράς ε, διατάξεων από τις αποφάσεις CTS e προς την οδηγία και έχουν κατατεθεί από ε, ευρωβουλευτές όλων των πολιτικών ομάδων και είναι πολύ σημαντικές γιατί συνδέονται με τις βασικές αρχές της οδηγίας, οργάνωση της αγοράς, δικαιώματα και υποχρεώσεις των ε, κατηγοριών των εμπορευομένων, ε, διαφάνεια και το καθεξής. Δεχόμαστε εμείς αυτή τη μεταφορά. Η πρόθεση του Κοινοβουλίου είναι να δώσει μεγαλύτερη έμφαση σε αυτά τα στοιχεία με την ενσωμάτωσή τους στο διατακτικό της οδηγίας να έχετε κατά νου ότι η Προεδρία του Συμβουλίου έχει καταθέσει συμβαστικό κείμενο που κινείται στην ίδια κατεύθυνση. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό θα γίνει τελικά, θα μεταφερθούν αυτές οι διατάξεις στο διατακτικό. Ωστόσο, υπάρχει ένα στοιχείο στις τροπολογίες του κυρίου Σαλίνη ε, με το οποίο δεν συμφωνούμε. Η εξαίρεση του, του συστήματος αυτόματης αναγνώρισης ε, των πινακίδων. Λέει ο κ. Σαλίνη ότι είναι χαμηλής αξιοπιστίας αυτό το σύστημα, όμως άλλοι ευρωβουλευτές ε, ε, διαφωνούν γιατί αυτή η τεχνολογία γίνεται το ένα και πιο σημαντική, ιδίως ό,τι αφορά τις πόλεις και θέλουμε να διατηρηθεί ως δυνατότητα. Τώρα, για το κατά πόσο η νομοθεσία μας θα είναι μελλοντοστραφής. Ε, έγινε μια συζήτηση για το ποια συχνότητα θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Σαφώς και θα ήταν καλό να είναι ταυτόσιμη η συχνότητα ή συμβατή με αυτή του ETS. Όμως ε, ακόμα αυτό δεν έχει ε, επιτευχθεί, γι' αυτό ε, προτείνουμε να μείνουμε στο 5,8 που είχαμε προτείνει αρχικά. Η δυνατότητα των επιλογικών έργων ήδη υφίσταται και αυτό είναι θέμα μεταφοράς μεταξύ απόφασης και οδηγίας, ούτε εδώ υπάρχει ζήτημα λοιπόν. Άλλη τροπολογία που έτυχε ευρεία στήριξη είναι η επέκταση του συστήματος και για την ανταλλαγή πληροφοριών για τους παραβάτες για να καλύψουμε και τα καθεστώτα αστικής ε, πρόσβασης, όπως και άλλα τα τέλη, όπως ε, ε, τα βινιέτ και ούτω καθεξής. Θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διασφαλίσει την επιβολή όλων αυτών των ε, συστημάτων και θεωρούμε ότι αυτή η τροπολογία είναι επικοδομητική. Κάποιοι πρότειναν στις τροπολογίες τα κράτη-μέλη όχι μόνο να είναι υποχρεωμένα να ανταλλάσσουν πληροφορίες για την ταυτότητα των παραβατών στα διόδια, αλλά και να παρέχουν συνδρομή το ένα προς το άλλο για την ανάκτηση των ε, ποσών και στα διόδια και στα πρόστιμα που δεν έχουν καταβληθεί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη το προβλέπει αυτό στην πρότασή της, αλλά θα μπορούσε να υπάρχει και ένα δεύτερο βήμα που ε, θα ληφθεί πέντε χρόνια μετά τη θέση ισχύ της οδηγίας. Κατανοούμε όμως ότι θέλετε να κινηθείτε πιο γρήγορα. Καλή είναι αυτή η ιδέα, Συμφωνούμε λοιπόν και με την άμεση ε, εφαρμογή αυτής της διάταξης. Ευχαριστούμε. Κύριε Σαλίνη, έχετε το λόγο. Ωραία. Όπως βλέπουμε υπάρχει συνένεση για την ανάγνωση της πινακίδας. Είναι τεχνικό το ζήτημα. Πρέπει να το λύσουμε γιατί νομίζω ότι και η Κομισιόν στην πρότασή της δεν περιλαμβάνει την ανάγνωση της πινακίδας μεταξύ των τεχνολογιών που, προβλέ... που προτείνονται σήμερα στο παράρτημα, αλλά αναφέρεται αλλού με διαφορετική διατύπωση στο κείμενο. Αλλά νομίζω ότι έχουμε μια σωστή βάση ώστε να αναζητήσουμε συνενέσεις και συγκλήσεις για αυτό το σημείο που θα μας επιτρέψει να έχουμε βεβαίως να τηρήσουμε σωστά τους στόχους της οδηγίας. Συμφωνώ και με την σύνοψη της Κομισιόν. Έκανα παρατηρήσεις συνάδελφοι για τις τεχνολογίες, αλλά να πω γενικά ότι είμαι βέβαιος ότι σύντομα θα βρούμε συμβασμός και θα ευοδοθεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Σαλήνη. Υπενθυμίζω ότι η ψηφοφορία θα γίνει στις 24 Μαΐου στις 9 το πρωί. Allez, nous passons tout de suite. Ωραία. Ας περάσουμε στο τελευταίο σημείο της πρωινής συνεδρίασης. Καλώ τον κύριο Αλμπέρτο Πρέτσι να έρθει να μας παρουσιάσει τη μελέτη για τον περίφημο δρόμο του μεταξιού. Allez-y, venez nous Ωραία, συνάδελφοι, υπενθυμίζω ότι ο δρόμος του μεταξιού ε, προσδιορίζει αυτούς τους ε, παλιούς εμπορικούς δρόμους, την εμπορική σύνδεση μεταξύ Ασίας, Ευρώπης ε, και πλέον μιλούμε και για την ε, Αφρική, περνώντας από την ε, Ρωσία, τη Λευκορωσία, τη Γερμανία, την ε, Γαλλία και είναι ιδιαίτερα φιλόδοξο γιατί έχουμε να κάνουμε και με τα δημοσιονομικά βέβαια, αλλά και για μια επένδυση της τάξης των 130 δις ευρώ. σε αυτό το δρόμο του μεταξύ όμως έχουμε λάβει υπόψη και αυτή την κλιματική μάχη. Είμαστε διατεθειμένοι σήμερα να συνεργαστούμε περαιτέρω με, τον, με έναν από τους μεγαλύτερους εμπορικούς μας εταίρους, την Κίνα. Όλα αυτά τα ζητήματα λοιπόν που θα εξετάσουμε σήμερα, σας δίνω το λόγο για να μας παρουσιάσετε τη μελέτη σας για 10 λεπτά για να μπορέσουμε να κάνουμε μετά τη συζήτηση. Κύριε Πρέτη, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχουμε πλέον μία πολύ σημαντική ε, μελέτη πολιτικής για που έγινε στην Κίνα για τη συνδεσιμότητα μεταξύ Ασίας και Ευρώπης με μεγάλο γεωγραφικό πεδίο ε, και αφορά 65 χώρες, 60% του παγκόσμιου ΑΕΠ και 30% του παγκόσμιου πληθυσμού. Η ανάλυση που κάναμε της ε, πρωτοβουλίας αυτής δείχνει ότι περιλαμβάνει ε, σημαντικό βαθμό επικοινωνίας δεν υπάρχει ξεκάθαρος ε, σχεδιασμός με προϋπολογισμό ή κατάλογο έργων και δεν έχει σαφή γεωγραφικά όρια. Φαίνεται ότι κυρίως αφορά τις ε, ε, σχέσεις πεμονωμένων χωρών με την Κίνα. Σε ό,τι αφορά τους στόχους BRI, η Κίνα αναφέρει ότι στόχοι της είναι η βελτίωση της ε, διεθνούς κατανόησης και συνεργασίας. Αυτό αφορά πέντε τομείς. Συντονισμός πολιτικής, οικοδόμηση δυναμικού, απελευθέρωση και διευκόλυνση των, ε, του εμπορίου και των επενδύσεων, οικονομική συνεργασία και ανταλλαγές μεταξύ λαών. Οι πιθανοί στόχοι της Κίνας ε, επικεντρώνονται στις εξαγωγές εξοπλισμού προϊόντων και το καθεξής, έλεγχος ε, της ε, αλυσίδας ε, των logistics, βελτίωση της οικονομικής σύγκλησης σε όλη την Κίνα, μηχανισμός για την αύξηση της χρήσης του εθνικού νομίσματος της Κίνας και δημιουργία εναλλακτικών οδών για τις εισαγωγές ενεργειακών πόρων. Σε ό,τι αφορά την συμμετοχή της ε, Κίνας σε αυτή την πρωτοβουλία, γίνεται μέσω δανεισμού από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και επενδύσεις στις ξένες επιχειρήσεις. Πάνω από 80 προγράμματα βλέπουμε ότι ε, λαμβάνουν χρηματοδοτική στήριξη από την Κίνα για όλους τους τρόπους μεταφοράς. Είναι εταίροι των Κινέζων Ιδίω ό,τι αφορά τις επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μιλούμε για τις μεταφορές. Απόκτηση μετοχών σε λιμένες, αεροδρόμια και σιδηροδρομικούς σταθμού. Υπάρχει μια συγκέντρωση επενδύσεων στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως στα Βαλκάνια, αλλά και στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, ενώ ε, σε ό,τι αφορά τους λιμένες, οι επενδύσεις ε, διοχετεύονται σε ολόκληρο το δίκτυο που συνδέει την ε, Ευρώπη με την Κίνα. Αυτή η συνεργασία μεταξύ Ασίας και Ευρώπης γίνεται σε τρία επίπεδα. Πρώτον, σε ό,τι αφορά το BRI, κυρίω η συνεργασία γίνεται μέσω διμερών συζητήσεων με μονομένα κράτη-μέλη και όχι με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. 20 κράτη-μέλη και 11 άλλες ευρωπαϊκές χώρες ε, υπέγραψαν από το 2014 και μετά μνημόνιο κατανόησης με την Κίνα. Υπάρχει συγκεκριμένο πλαίσιο συνεργασίας με την Κίνα στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, το πλαίσιο 16 1, που έχει χρησιμεύσει ως ε, πλατφόρμα ανακοίνωσης του BRI. 11 κράτη-μέλη, 5 ευρωπαϊκές χώρες στην Κίνα και τέλος, ε, εμείς ε, προάγουμε την πλατφόρμα διασύνδεσης για να, σε ό,τι αφορά τις ε, επενδύσεις της Κίνας σε όλο το δίκτυο διασύνδεσης με την Κίνα για τον BRI. Θεωρούμε ότι ακόμα υπάρχει αβεβαιότητα βέβαια. Επενδύσεις στη, στο νέο δρόμο του μεταξύ είναι μόνο μικρό τμήμα των γενικών επενδύσεων που θα λάβουν χώρα, ανεξάρτητα από τον BRI. Δεύτερον, είναι πολύ δύσκολο να προδικάσουμε το αποτέλεσμα. Από την μελέτη αναλύουμε τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ ε, Κίνας και Ευρώπης. Αυτή τη στιγμή, αλλά και στο μέλλον, το εμπόριο είναι κυρίως διαθαλάσσεις. Θεωρούμε ότι το BRI ενδεχομένως ε, να ωφελήσει τους λιμένες της Νοτιού Ευρώπης και ταυτόχρονα θα υπάρξει μια μετατόπιση προς ε, τις συνδρομικές μεταφορές έως 3.000 ε, BTUs μέχρι το 2040. Σε ό,τι αφορά τώρα τις ευκαιρίες που προσφέρει το BRI οι Κινέζοι είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν ε, ρίσκα και να οικοδομήσουν και να επενδύσουν σε οικοδομικά έργα. Θέλουν να επενδύσουν και ε, στις αερογραμμές και στο σιδηρόδρομο. 50-60 παραπάνω τρένα σε κάθε κατεύθυνση μέχρι το 2040 νομίζουμε θα υπάρχουν. Εάν αυτό είναι οικονομικά βιώσιμο, οι υπηρεσίες θα είναι επωφελείς για την ευρωπαϊκή βιομηχανία και κυρίως αυτό συνδέεται με την εξισορρόπηση των ροών μεταξύ Ανατολής και Δύσης, δηλαδή να αυξήσουμε τις εξαγωγές μας προς ε, την Κίνα και έτσι να αυξήσουμε τους εξαγωγείς μας. Ταυτόχρονα, το BRI έχει και προκλήσεις. Πρώτον, ε, οι Κινέζοι έχουν ε, την κυριότητα της αλυσίδας ε, των logistics και αυτό μπορεί να αυξήσει την, το μερίδιο της αγοράς τους. Δεύτερον, τα τεχνικά πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μη ευρωπαϊκές χώρες μπορούν να επανομευθούν από την προώθηση ε, διαφορετικών τεχνικών προτύπων. Τρίτον, τα προγράμματα υποδομών μπορούν να εφαρμοστούν γιατί υπάρχει διαθέσιμη κινέζικη χρηματοδότηση με λιγότερο σημείο εστίαση σε την βιωσιμότητα ή τη ζήτηση των υπηρεσιών που υποτίθεται ότι θα καλύψουν οι υποδομές μεταφορών. Μετά υπάρχει έλλειψη ξεκάθαρου σχεδιασμού BRI και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αλληλεπικαλύψεις με άλλα εντός ή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τέλος, σημαντικές προκλήσεις στους τομείς της αμοιβαιότητας σε ό,τι την πρόσβαση στους, ε, στα δημόσια έργα και ίσο παιδί του αγωνισμού ε, στις εξεγωγές. Σε ό,τι φορά τώρα την ε, ετοιμότητα του ευρωπαϊκού συστήματος, θεωρούμε ότι ο ευρωπαϊκός διάδρομος που κατά πιθανότητα θα ε, επηρεαστεί είναι το δίκτυο της Βόρειας Θάλασσας και της Βαλτικής. Αλλά δεν είναι σαφές αυτή τη στιγμή εάν και κατά πόσο και πού ε, η κίνηση BRI θα οδηγήσει σε συμφόρηση. Η μελέτη δείχνει λοιπόν ότι δεν έχουμε επαρκή στοιχεία για να προτείνουμε στην Επιτροπή τροποποιήσεις ε, του προγράμματος εξαιτία του BRI. Τέλος, σε ό,τι αφορά τις συστάσεις. Πρώτα απ' όλα θέλουμε να διατηρήσουμε το διάλογο και τη συνεργασία με την Κίνα θέλουμε μεγαλύτερη σαφήνεια για τους μελλοντικούς σχεδιασμούς υπό το BRI και να ενισχύσουμε τις ε, εργασίες της πλατφόρμας σύνδεσης και συνδεσιμότητας. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά την προστασία των ευρωπαϊκών συμφερόντων, θέλουμε να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την ε, πρόοδο ε, υπό την ολοκληρωμένη συμφωνία περί επενδύσεων, να διασφαλίσουμε ότι το ERTMS παραμένει το κατεξοχήν πρότυπο εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως συμβαίνει αυτή τη στιγμή και στην Ασία, να διασφαλίσουμε την αμοιβαιότητα πρόσβασης στις ε, αγορές δημοσίων έργων και να αναπτύξουμε ένα εργαλείο βάσει της ε, πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να διασφαλίσουμε πλαίσιο για να ελέγχουμε ε, τις άμεσες ξένες επενδύσεις, να ενθαρρύνουμε την Κίνα να συμμετάσχει στις κριτήριες γραμμές του ΟΣΑ για, τις, ε, για τα export credits και τέλος να εισαγάγουμε περιοδικές αναθεωρήσεις των ε, επιρροών του BRI στο TEN-T. Ιδίως στο πλαίσιο της πλατφόρμας συνδεσιμότητας για, για τα συγκεκριμένα διαδρόμους TNT και BRI ξεκινώντας από τη σύνδεση μεταξύ ε, του, του διαδρόμου βασικού δικτύου ε, Βόρειας Θάλασσας Βαλτικής και του διαδρόμου που βγαίνει από Κίνα, Καζακστάν, Λεύκο Ρωσία, Πολωνία, Γερμανία και κατοχώς. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρέτη για την παρουσίαση του θέματος. Να αρχίσουμε μέσω τη συζήτηση για το θέμα αυτό βέβαια, για τον δρόμο του μεταξιού και πρώτος ο κύριος Βαντεκάμπ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρέπει να σας πω ότι ευχαριστώ πολύ τον κύριο Πέτρη ε, για αυτή την μελέτη. Είμαι και μέλος της αντιπροσωπείας για την Κίνα. Αυτό που λέγαμε παλιότερα Όμπερ και τώρα λέγεται BRI είναι ένα σημείο το οποίο πολύ συχνά βρίσκεται στην ορίστη διάταξη. Και ε, η μελέτη αυτή περιέχει πολύ σημαντικές πληροφορίες και διαρωτώ με, κυρία Πρόεδρε, μήπως και στην Επιτροπή ΑΦΕΤ ε, πρέπει να συζητηθεί αυτή η μελέτη. Γιατί πρόκειται για πολύ σημαντικά γεωπολιτικά ζητήματα που κατά τη γνώμη μου θα πρέπει και η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου να τα εξετάσει. Αυτό που είναι σημαντικό σε, με τις, ε, σε ό,τι αφορά τις σχέσεις μας ε, με την Κίνα ε, και πιο συγκεκριμένα εδώ έχουμε να κάνουμε με τις μεταφορές. Η συστάση της σελίδα 18 που διάβασα σήμερα το πρωί ως ήθιστα είναι ιδιαίτερα ευγενικά διατυπωμένες και με μεγάλη προσοχή. Ε, ως προς το τι πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή. Για να είμαι ειλικρινής, όταν κανείς ε, συνομιλεί με τους ε, Κινέζους συναδέλφους, πάντα γελούν, πάντα χαμογελούν, είναι πολύ φιλικοί και πάντα θέλουν να υπάρχει πολύ καλή συνεργασία με την Ευρώπη, αλλά κάποιες φορές είναι και μια μορφή απεικιοκρατίας. Συγγνώμη που χρησιμοποιώ αυτό τον όρο, αλλά αν δείτε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή με τα ποσά που επενδύει η Κίνα και τα όσα συζητήσαμε χθε ε, το μεσημέρι για το ΣΕΦ, εμείς τι είμαστε πιόνια ε, σε όλη αυτή την ιστορία. Και τι θέλει τελικά η Ευρωπαϊκή Ένωση μακροπρόθεσμα. Ο κύριος Πρέτη είπε πολύ σωστά ότι η Κίνα δεν ε, συνομιλεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά με τα επιμέρους κράτη-μέλη και πιο συγκεκριμένα στην Ανατολική Ευρώπη. Αν δείτε τον κατάλογο των έργων που χρηματοδοτεί η Κίνα στην Ανατολική Ευρώπη, αλλά και στην πόλη μου, στο Ρότερνταμ όπου έχουν αγοράσει ε, τμήμα του τερματικού σταθμού. Τότε μπορώ να θέσω το εξή ερώτημα στον κύριο Πρέτη. Τι πρέπει να κάνουμε από εδώ και πέρα. Γιατί μπορούμε να συνεχίσουμε να είμαστε ευγενικοί, αλλά οι ε, είναι τεράστιε, κινούνται πολύ γρήγορα οι Κινέζοι και πρέπει να δούμε κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να τα βγάλει πέρα σε ό,τι αφορά τον BRI που μας παρουσιάζει συνεχώς η γενεστική πλευρά, βέβαια με το χαμόγελο στα χείλη. Δύο τεχνικά ερωτήματα. Σε ό,τι φορά την, ε, τη, συσχέτιση μεταξύ ε, της επενδυτικής τράπεζας υποδομών στην Ασία και της NDB. Δεν θυμάμαι τώρα τι είναι αυτό, αλλά θα σας το βρω. Η νέα αναπτυξιακή τράπεζα της Κίνας είναι αυτή. Ε, είναι σωστή η εντύπωσή μου ότι αυτή η τράπεζα είναι πολύ μεγαλύτερη ε, και έχει πολύ μεγαλύτερη διδημιδιωτική ικανότητα από ότι η Ασιατική Τράπεζα Επενδύσεων στον τομέα των υποδομών. Και ένα άλλο σημαντικό στοιχείο της έκθεσης είναι ότι η Ευρώπη αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα με το ERTMS, ε, κατέχει ηγετική θέση σε ό,τι αφορά τα παγκόσμια πρότυπα. Μπορούμε να τη διατηρήσουμε αυτή τη θέση ε, μακροπρόθεσμα, λαμβάνοντας υπόψη τη στάση της Κίνας. Ε, τέλος, τα όσα συζητήσαμε πριν από δύο εβδομάδες για τον τουρισμό. Ποια είναι η αμοιβαιότητα. Εμείς ακόμα δεν μπορούμε να επενδύσουμε στην Κίνα, πάνω από 50%. Και δεν θέλω να σπείρω τον πανικό, αλλά αν διαβάσει κανείς αυτή την μελέτη με τις τεράστιες επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων, εκατομμυρίων και εμείς έχουμε ένα σεφ 33 δις. Σιγά τα ΟΑ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ αγαπητέ Βαντεκάμπ κύριε Ερτούγκ. Και από τη δική μου λοιπόν πλευρά και τη δική μου πολιτική ομάδα ένα θερμό ευχαριστώ για την ενδιαφέρουσα εκθέση και μελέτη. Πράγματι, τώρα πώς να το πω, η Ευρωπαϊκή Ένωση ίσως έχει ένα μειονέκτημα με την έννοια ότι είμαστε ένωση κρατών και δεν είμαστε οι Ηνωμένε Πολιτείες της Ευρώπης ας πούμε. Και αυτό φαίνεται καθαρά στο γεγονός ότι οι 28 χώρες μέλη αντιμετωπίζουν με διαφορετικό τρόπο το θέμα. Υπάρχουν χώρες μέλη οι οποίες ενδιαφέρονται πολύ στη συνεργασία, για τη συνεργασία αυτή, διότι παράγεται και πλούτος και αυτό τους ενδιαφέρει και υπάρχουν και χώρες μέλη που τα βλέπουν αυτά τα πράγματα διαφορετικά ή εν πάση περιπτώσει ενδέχεται και να μην έχουν αντιληφθεί τη σημασία του εγχείρηματος. Αν η Κίνα είχε διαφορετική κρατική μορφή και συνταγματικό χαρακτήρα, τότε ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Πάντω, θεωρώ ότι θα πρέπει να διαγνώσουμε τις προτεραιότητες και να αντιδράσουμε αναλόγως. Όταν μιλούμε για τη νέα οδό τη μετάξη, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι πρόκειται για δύο κέντρα, ίσως και τέσσερα εξουσία: Κίνα, Ρωσία, Κεντρική Ασία και Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για τους τέσσερις μεγάλους φορείς που θα πρέπει να προσπαθήσουμε να τους βάλουμε να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι. Εγώ είμαι μέλος της αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με την Κεντρική Ασία και υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τις χώρες της Κεντροασιατικής Συνεργασίας για συνεργασία, χώρες με τις οποίες οι εμπορικές μας σχέσεις είναι πολύ χαμηλά. Θα μου πείτε βέβαια υπάρχουν θέματα ανθρώπινων δικαιωμάτων κλπ. Σωστό είναι αυτό. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα πρέπει να αποφύγουμε να συνεργαστούμε μαζί τους. Θεωρώ ότι μπορούμε να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία αυτή με την δημιουργία αυτής της σύνδεσης που έχει πραγματικά παγκόσμιες διαστάσεις και έχει και πολύ ενδιαφέρον, για παράδειγμα, στη σελίδα 22 της μελέτης, οι διάφοροι οικονομικοί διάδρομοι τους οποίους περιλαμβάνετε εσείς. Δύο από αυτούς, China, ε, Russia, Mongolia και ο άλλος που αποτελούν την σύνδεση και προς εμάς εδώ στην Ευρώπη. Και νομίζω ότι εδώ δεν πρέπει να απευθυνθούμε μονάχα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Υπηρού, διότι υπάρχουν και χώρες οι οποίες δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βρίσκονται όμως καθοδόν αυτής της ε, οδού της μετάξης. Εν τέλει πάντως, το ρόλο δεν θα παίξουν μονάχα τα χρήματα, πολύ σωστά το είπε ο κ. Βαντεκάμπ, αλλά και η πολιτική βούληση θα παίξει κεντρικό ρόλο εάν και κατά πόσον δηλαδή θέλουμε και εμείς να υποστηρίξουμε, να συνδιαμορφώσουμε αυτό το σχέδιο μαμούθ. Γι' αυτό θα προτείνω. Ακούστηκε βεβαίως και η Επιτροπή Εξωτερικών, ΑΦΕΤ, αλλά και η αντιπροσωπεία για τη σχέση με την Κεντρική Ασία. Και να προσκαλούνται και μέλη από αυτήν, την αντιπροσωπική δική Ασία, από την Επιτροπή Εξωτερικών κλπ. Και σωστό θα είναι βέβαια οι χώρε μέλη να προσπαθήσουν να ακολουθήσουν μια νέα πορεία. Πάντω, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εν προκειμένου πιο συγκεκριμένα η Επιτροπή μα μπορεί να δώσει μια πρώτη όθηση. Διότι έχουμε συζητήσει ήδη πολύ για το θέμα αυτό, αλλά λίγα πράγματα έχουν γίνει συγκεκριμένα. Ευχαριστώ κύριε Ερτούκ. Ο κύριος Τελίτσκα. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και τον κύριο Πρέτη για τη μελέτη. Σημαντική πρωτοβουλία, παρέχει πολλές πληροφορίε και έρχεται και στη σωστή στιγμή. Λέχθηκε ήδη τη μεγάλη στρατηγική σημασία έχει το εγχείρημα αυτό. Ωστόσο, ας μην γελιόμαστε λίγη επιρροή μπορούμε να ασκήσουμε στο εάν οι Κινέζοι θα προχωρήσουν με πλήρη ταχύτητα ή όχι. Κατά πάσα πιθανότητα έτσι θα προχωρήσουν, δηλαδή έχουν ε, ένα στρατηγικό γεωπολιτικό στόχο στο μυαλό τους και αυτόν θα ακολουθήσουν. Και μάλιστα από τα ύψιστα ε, επίπεδα της πολιτικής τους ιεραρχίας. Καμιά φορά μιλούμε για τις ελλείψεις του στρατηγικού σχεδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά την εξωτερική συνδεσιμότητα. αν δούμε δηλαδή τα ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου ακόμα έχουμε όλα αυτά τα ε, προβλήματα. Ακόμα δεν είμαστε αφεντικά της μοίρας μας στα θέματα αυτά. Και πάλι ας μην γελιόμαστε. Εάν γίνει αυτή η γραμμή αυτή, ποιος θα την λειτουργεί, με ποιες προϋποθέσεις, με ποια πρότυπα. Και πάλι η δική μας δυνατότητα επιρροής μπορεί ίσως να είναι σημαντική, αλλά δεν θα είναι δεν θα είναι καθοριστική, θα είναι το πολύ περιθωριακή. Ας φανούμε λοιπόν, ας αναλάβουμε δράση ταχύτερα. Με ορισμένα από τα σχόλια συμφωνώ. Αν θυμάμαι καλά όμως κύριε Πρέτη, είπατε ότι θα πρέπει να αναλύουμε σταδιακά την κατάσταση. Όμως ίσως να είναι άβολες οι αναλύσεις αυτές τα αποτελέσματά τους. Χρειαζόμαστε, χρειαζόμαστε περισσότερο ενεργή δράση. Χρειαζόμαστε μια κοινή πολιτική μεταφορών ή κοινή πολιτική εξωτερικών μεταφορών. Εγώ θα έλεγα να αρχίσουμε ήδη από τα ε, έργα των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών που όλα αυτά γίνονται στη βάση κάποιας μελέτης σκοπιμότητας, για παράδειγμα, του Βόρειου Διαδρόμου. Θυμάμαι το περιεχόμενο της μελέτης σκοπιμότητας που βασιζόταν σε υποθετικές εξελίξεις κάποιου εμπορίου που θα έρχεται από την Κίνα μέσω Καζακστάν. Να επανεξετάσουμε αυτές τις μελέτες σκοπιμότητας και να δούμε εάν εφαρμοστούν Πώ ακριβώς, αν τα πράγματα αυτά που βλέπουμε τώρα εφαρμοστούν, πώ θα αλλάξει το περιεχόμενο της μελέτη σκοπιμότητας, διότι έχουμε ήδη επενδύσει δισεκατομμύρια και θα επενδύσουμε και άλλα. Αυτό θα μα δείξει τι είδου επιπτώσει έχουν αυτέ οι κινήσει. Εάν τα φορτία θα έρχονται από την Κίνα μέσω Καζακστάν και την Κεντρική Ασία, το χρήμα παίζει τον βασικό ρόλο. Είναι τόσο εύκολο λοιπόν να μετακινηθεί το φορτίο από τη διαδρομή Α στη διαδρομή Β. Και ανεξαρτήτως τώρα της ποιότητας της μελέτης που είναι καλή και των συμπερασμάτων που προσφέρουν τροφή για σκέψη, εδώ το βασικό θέμα είναι να φτάσουμε σε μια κοινή πολιτική μεταφορών. Πέραν των ορίων της Ένωσης. Και για την ώρα, εγώ τέλος πάντων είμαι από μια χώρα η οποία ατυχώς στο υψηλότερο πολιτικό επίπεδο κάνει business με την Κίνα και μερικοί και ο Τσέχος πρόεδρος κάνουν τέτοια πράγματα. Το βασικό μήνυμα λοιπόν πρέπει να προέλθει από την δική μας Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο είναι αν θέλουμε να αποφύγουμε να αποκοπεί ένα μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να υπάρξουν αρνητικές συνέπειες χρειαζόμαστε μια κοινή πολιτική με ξεκάθαρη στρατηγική και με εναλλακτικέ επιλογέ και βέβαια δεν είμαι αφελή να αναμένω ότι θα πετύχουμε τίποτε άλλο παρά περιορισμό των ζημιών. Να μην πω σε λεπτομέρειε, ελπίζω ότι θα έχουμε περισσότερο χρόνο κάποια στιγμή στο μέλλον να συζητήσουμε περισσότερε λεπτομέρειε στην βάση ποιον, πιο συγκεκριμένων ωστόσο στοιχείων που θα μα δώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ η κυρία Ντεμόντε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ για αυτή την ενδιαφέρουσα μελέτη. Έγκαιρη για την Επιτροπή μας, αλλά κάπως λιγότερο για την Κομισιόν, προς την οποία είχα απευθύνει μια ερώτηση τον Οκτώβριο 16 σχετικά με διάφορους ε, Ευρωπαίους, ευρωπαϊκούς λιμένες, ρωτώντας δηλαδή τη μελέτη αντικτύπου είχε κάνει η Κομισιόν για τους λιμένες αυτούς. Σε σχέση όχι μόνο με τη στρατηγική του σημασία, αλλά και σε σχέση επίσης με τις επενδύσεις, τα δικαιώματα των εργαζομένων κλπ. Και είχα μια ανελειπή, συγγνώμη, μια απάντηση εκ μέρους της ε, Κομισιόν, που μιλούσε μόνο για κάποιους ελέγχους από το κράτος. Εντάξει, αλλά εδώ θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με την παρουσία των Κινέζων. Γιατί έχουμε αύξηση του πληθυσμού και δεν μπορούμε να απαντάμε ότι οι πρώτες και η διακίνησή τους θα πρέπει να προσεγγίζονται μόνο από, εμπορικό, από εμπορική σκοπιά. Θα πρέπει λοιπόν να πούμε τι γίνεται με την προσπάθεια ελέγχου κόμβων επιμελητίας και νομίζω θα πρέπει να υπάρχει πάντα μια αναλλακτική και ιδιαίτερα στην ε, περίπτωση των Βαλκανίων θα πρέπει να αναζητήσουμε άλλες διόδους γιατί η θαλάσσια, ο θαλάσσιος διάδρομος όπως το είσατε και εσείς είναι αυτός που υπερισχύει και αυτό αφορά την, τη δυνατότητα μεταφοράς αλλά και την εξάλληψη φραγμών. Εντάξει, για τα Βαλκάνια η Κίνα αναζητεί μια εναλλακτική, δηλαδή να μην έχει μόνο μία οδό μεταφορών, αλλά αναζητούν εναλλακτικέ για να μην ε, έχουν αποκλειστική σύνδεση και σχέση με χώρες μέλη. Οπότε θα ήθελα να ρωτήσω αν, μπορούμε να, αν θα μπορούσαμε να έχουμε και μια αντίστοιχη μελέτη, δηλαδή μια μελέτη αντικτύπου για να δούμε ακριβώς τι εναλλακτικέ υπάρχουν, μόνο για τις εξαγωγές που ενδιαφέρουν την Κίνα, αλλά και για τα συμφέροντα της Ευρώπης, να δούμε δηλαδή τι δυνατότητες υπάρχουν, ώστε να είμαστε και ενεργοί παράγοντες, πρωταγωνιστές, ώστε να είμαστε και εξαγωγείς. Και δεύτερη ερώτηση. Γνωρίζουμε κατά πόσο σήμερα υπάρχουν αυτούσιες επενδύσεις και χρηματοδοτήσεις, δηλαδή κατά κάποιο τρόπο πώς σχετιζόμαστε άμεσα οικονομικά με την Κίνα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Τιμοντέο, κύριο. Ε, Ρικέ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Χαίρομαι που ο κύριος ε, Βαντεκάμπ ε, έλαβε το λόγο προηγουμένως και είπε αυτά που είπε με μέτρο. Ναι, όντως πρέπει να έχουμε νου τις διεθνείς σχέσεις, την συνένεση, τη συνεργασία, τη διεθνή και την βελτίωση της ε, παγκόσμιας ευημερίας. Βέβαια, για αυτά τα θέματα υπάρχει κάποια ανησυχία. Καταρχάς, επειδή έχουμε να κάνουμε μια αυταρχική δύναμη με κεντρικό σύστημα εξουσίας και επιχειρήν το οποίο διαχειρίζεται αυτή η κεντρική εξουσία και είδαμε επίσης σε σχέση με τους συνομιλητές ότι η Κίνα συνομιλεί με τις χώρες ως εταίρους ώστε να κατακαιρματίσει την νότα που υπάρχει ιδιαίτερα στην Ευρώπη. Και στην Ευρώπη απευθύνεται στους πιο αδύναμους κρίκους στο σύστημα μεταφορών η Κίνα. Δεύτερη παρατήρηση για τις ανταλλαγές τις χρηματοοικονομικές. Για την Κίνα είναι πιο ενισχυτικό αυτό. Και ποσοτικά και ποιοτικά αλλά και χρηματοοικονομικά. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι υπάρχει δυνατότητα ελέγχου ή παρεμπόδισης αυτού του βήματος που κάνει η Κίνα σε σχέση με αυτές τις χώρες. Αλλά εκτός και να στείλουμε στρατούς, νομίζω θα πρέπει να, δούμε τι θα κάνουμε οικονομικά, να αντιδράσουμε οικονομικά σε επίπεδο, σε επίπεδο ανταλλαγών. Γιατί όντως υπάρχει μια στάση νέο απεικιοκρατική εκ μέρους της Κίνας. Και με ανησυχεί η αδύναμη αντίδραση της Ευρώπης αλλά και η εσωτερική συζήτηση που γίνεται στο εσωτερικό της μεταξύ χωρών μελών. Αν δείτε αυτά που προτείνονται στο χάρτη, θα δούμε ότι υπάρχουν συγκεκριμένα γεωστρατηγικά συμφέροντα όσον αφορά την προσεγγίση της Κίνας και βαθμία ο οικονομικός και οργανωτικός έλεγχος της επιμελητίας και των οδών της ε, έρχεται σε κινέζικα χέρια. Αν μου λοιπόν τι γίνεται και στην Αφρική, υπάρχουν λόγια ανησυχία. Πάντως εγώ νομίζω ότι το BRI είναι μια απεικιοκρατική προσέγγιση υπέρ της Κίνας και βεβαίως αυτό αφορά και εσωτερικές διαμάχες μεταξύ των χωρών μελών. Και όσον αφορά την επιμελητία και τις μεταφορές, η τεχνική που εφάρμοσαν αφορούσε τις ε, ανταλλαγές και την ε, προστασία μηχανικών μυστικών να πω και κάτι άλλο. Τι άποψη έχετε για την οδό της Αρκτικής του Βορρά. Πώς θα επηρεάσει βραχυπρόθεσμα αλλά και αργότερα τα εγχειρήματα τα κινέζικα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ρικέ, κύριε Νταλούντε. Έχετε το λόγο εσείς. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά που ακούσαμε. και μας αποδεικνύουν ότι υπάρχει εδώ ένα σημαντικό δυναμικό, δηλαδή μπορούν να δημιουργηθούν υποδομές, σιδηροδρομικές και άλλες ως εναλλακτικές μορφές μεταφορών. Το εμπόριο μεταξύ Ευρώπης και Κίνας μέχρι το 2020 θα αυξηθεί σημαντικά με σημαντικά ποσοστά. Οπότε θα πρέπει να αναζητήσουμε βιώσιμε λύσει. Ταυτόχρονα υπάρχει ένα κίνδυνο. Αν αφήσουμε την Κίνα να χρηματοδοτήσει αυτέ τι υποδομέ, τότε θα πρέπει να σκεφτούμε σοβαρά τι επιπτώσει από την κυριαρχία τη Κίνα σε αυτέ τι ε, υποδομέ σε σχέση πάντοτε με το παγκόσμιο εμπόριο. Θα πρέπει να μελετήσουμε καλύτερα τις γεωπολιτικές επιπτώσεις αυτών των εξελίξεων και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να επικεντρωθούμε στην έκθεση του κύριου Βαντακάμπ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πάμε στο Ευχαριστώ για αυτή την ταυμάσια ε, εισηγήση, χρήσιμη και κέρια για αυτά που ζούμε και την περσμένη εβδομάδα είχαμε συζητήσει στο Στρασβούργο τις ε, εξαγγελίες Τραμπ σε σχέση με τις αγωγές αλουμινίου και στην Ένωση είπαμε ότι μας ανησυχεί αυτός ο αθέμητος ανταγωνισμός σε αυτές τις αγορές εκ μέρους της Κίνας που επηρεάζει σημαντικά και το τομέα των μεταφορών. Οπότε θα πρέπει πέρα από αυτά που λέμε εμείς εδώ να πάμε παραπέρα στις δράσεις μας ως Ένωση, η Κομισιόν, εμείς ως νομοθέτης γιατί θα πρέπει ως Ένωση να αντιδράσουμε, όχι μόνο με μονομένα ως χωρές μέλη, γιατί θα πρέπει να αποτιμήσουμε τις επιπτώσεις στη μηχανία μας, του δρομικές μας εταιρείες κλπ. Τομείς που θίγονται από τον ισχυρό ανταγωνισμό της Κίνας στην Ένωση. Θα μπορείτε να μας πείτε τι γίνεται με την ε, γραμμή υψηλής ταχύτητας τη συνδρομική μεταξύ Βουδαπέστης και Βουκουρεστίου και την εμπλοκή της Κίνας και πώς θα μπορούσαμε να προσπίσουμε τα συμφέροντα των Ευρωπαίων Βιομηχανιών, των Ευρωπαϊκών Βιομηχανιών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Λαϊκή Πρόεδρος. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει μια προεκβολή χρηματοοικονομική. Ένα τρεις, ένα τρεις ευρώ έχει ήδη ανακοινώσει η Κίνα και έχουν ξεκινήσει αυτές οι εργασίες. Έχουν αρχίσει τα εργοτάξια. Σήμερα έχουμε 60 χώρες που έχουν συνδεθεί, 260 έργα που έχουν υπογραφεί και ο κύριος Στενίσκα και ο κύριος Ρικέ και ο κύριος Φοντεκάμπ Το ανέφεραν ότι η κύρια εδώ ανησυχία των Ευρωπαίων είναι καταρχάς για θέματα διαφάνειας που αφορούν τις αγορές, κανόνες κοινωνική, περιβαλλοντική κλπ. Και δεύτερο, κατά πόσο αυτά τα έργα είναι έργα τα οποία θα ωφελήσουν τη Δυτική Ευρώπη. Και εδώ τίθεται ένα απλό ερώτημα. Σήμερα η Κίνα είναι έτοιμη να προβεί σε μια παγκόσμια διακυβέρνηση. Εγώ λέω όχι. Οπότε το πραγματικό ερώτημα είναι κατά πόσο αυτά τα έργα ανταποκρίνονται στις προσδοκίες της των Ευρωπαίων πολιτών. Όχι θα έλεγα. Μετά δεύτερο ερώτημα είναι ποιες είναι οι επιπτώσεις αυτών των έργων προς τους, σε σχέση με τους δικούς μας στόχους κλιματική αλλαγή και δρόμος του μεταξύ. Ωραία, θαυμάσια αυτά που λέμε για το σιδηρόδρομο. Αν δούμε όμω την ίδια την φύση αυτών των έργων υποδομή, θα δούμε ότι αναπόφευκτα οδηγούν σε υπερβάσεις κόστους, αφενός, σε υπερδιαστασιολογήσεις και περιτά κόστη, με τεράστιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Οπότε, εγώ έχω δύο απλές ερωτήσεις. Σήμερα η Ευρώπη μπορεί να προβάλλει αυτές τις ανησυχίες καταρχάς σε σχέση με τη διαφάνεια στις αγορές και στην τήρηση στα πλαίσια των διαγωνισμών κανόνων κοινωνικών και περιβαλλοντικών και δεύτερον μπορούμε να φτάσουμε σε μια παγκόσμια διακυβέρνηση γιατί ξέρουμε σε αυτήν την περίπτωση ο ηγέτης θα είναι η Κίνα. Et donc vous avez... Οπότε... Α. Κύριε Πρέτα, έχετε το λόγο για να απαντήσετε. Καλή τύχη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σε ό,τι αφορά το πρώτο σύνολο ερωτήσεων, η τράπεζα NDB η Αναπτυξιακή Τράπεζα της Κίνας. Σαφώς και ε, συμμετέχει σε αυτό. Περίπου 110 δις δολάρια ε, σε πιστώσεις που αφορούν και την Κίνα αλλά και τη Βραζιλία, τη Ρωσία και την Νότια Αφρική. Στα πρώτα στάδια ανάπτυξης του BRI ήταν περισσότερο επενδυτικές τράπεζες, εμπορικές τράπεζες της Κίνας. Τώρα, τα τελευταία χρόνια βλέπουμε μια αύξηση της χρηματοδότησης και από άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, η Asian Infrastructure Investment Bank και η Νέα Αναπτυξιακή Τράπεζα. Δεύτερον, κατά πόσο το ERTMS θα παραμένει το πρότυπο. Η μελέτη δεν εξέτασε το μέλλον του ERMTS. Μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα πρότυπο αυτή τη στιγμή και είδαμε ότι χρησιμοποιείται ευρέως και στην Ασία. Αλλά δεν μπορούμε να προκαταβάλουμε ότι θα είναι το ίδιο αυτό στο μέλλον. για τις παρατηρήσεις που κάνατε προηγουμένως. Νομίζω ότι προκύπτουν και στα συμπεράσματα Δηλαδή θα πρέπει να επικεντρωθούμε στη διασύνδεση με τα ευρωπαϊκά μεταφορικά συστήματα. Πέραν των ζητημάτων που δεν συνδέονται με τις μεταφορές, αμοιβότητα δηλαδή στην πρόσβαση ε, στην αγορά των δημοσίων έργων και στις εξαγωγές. για τις εξαγωγές και την αξιολόγηση αντικτύπου και τους οικονομικούς δεσμούς με την Κίνα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση του αντικτύπου των κινέζικων επενδυτικών ε, προγραμμάτων υποδομών στην Ευρώπη σίγουρα θα ήταν κάτι το χρήσιμο. Μπορεί να γίνει και κατά τη γνώμη μου απαιτεί ένα πιο συγκεκριμένο σημείο εστίαση σε συγκεκριμένα προγράμματα υποδομών σε σχέση με τον αντίκτυπό τους. Γιατί το BRI είναι ιδιαίτερα ευρύ. Από τεχνική άποψη λοιπόν είναι δύσκολο να εκτιμήσει κανείς το συνολικό αντίκτυπο σε πολλούς ε, τομείς. Μεταφορές, απασχόληση, εμπόριο και το καθεξής που συνδέονται με το BRI για τις ευκαιρίες που προκύπτουν για τις ευρωπαϊκές εξαγωγές. Αυτό εξαρτάται από πολλούς ε, παράγοντες. Αυτή τη στιγμή μπορούμε να πούμε ότι έχουμε σημαντικές ε, ευρωπαϊκές εξαγωγές προς την Άπο Πριν ανέφερα κάποια 60 εκατομμύρια TUs. Αυτό δείχνει ότι ήδη οι ευρωπαϊκές ε, επιχειρήσεις εξάγουν προς την Άπο Ανατολή, σαφώς ε, και εντοπίζει έκθεση δυνατότητες αύξησης αυτών των ροών. Οι υποδομές, μεταφορές ε, και επιμελητίας, καθώς και οι υπηρεσίες, κατά τη γνώμη μας, είναι κινητήριος μοχλός αύξησης αυτών των εξαγωγών. Όχι μόνο για τις ευρωπαϊκές υποδομές, αλλά και για τις χώρες ε, διαμετακόμισης. Υποδομές δηλαδή και στην Κεντρική Ασία. Σε ό,τι αφορά τους οικονομικούς δεσμούς ε, με την Κίνα, κατά τη γνώμη μας ήδη έχουμε πολλούς τέτοιους οικονομικούς δεσμούς, αλλά αυτό συνέβαινε και προηγουμένως, πριν από την εκκίνηση του BRI του 2013 για παράδειγμα, επισκευή ορισμένων λιμένων στον Βασίλειο τη δεκαετία του 1990. Η αγορά του λιμανιού του Πειραιά που ξεκίνησε πριν από την επίσημη κίνηση του PRI. Από τεχνική άποψη λοιπόν νομίζω ότι ήδη υπάρχουν ε, ξεκάθαρη, ξεκάθαρα σημάδια ε, κινέζικων επενδύσεων στην Ευρώπη. Για την ε, οδό της Αρκτικής, για να είμαι ειλικρινής, δεν διερευνήσαμε το ζήτημα. Σαφώς και μπορούμε να το μελετήσουμε περαιτέρω στο μέλλον, αλλά δεν μπορώ να αποφανθώ αυτή τη στιγμή, γιατί δεν το έχουμε διερευνήσει συγκεκριμένα. Για την υπερταχεία στα Βαλκάνια, Αναφερθήκατε στην ε, οδό μεταξύ και τη σύνδεση μεταξύ Βουδαπέστης και Βουκουρεστίου. Είδαμε ότι έχει υπάρξει επένδυση. Βάσει τη αναθεώρηση βιβλιογραφία, είδαμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέτασε το ζήτημα τη συμμόρφωση με του ευρωπαϊκού διαγωνισμού μέχρι το 2017 που παραδόθηκε η μελέτη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπάρχει συμβαλόμενο μέρος, μία επιχείρηση ε, η οποία ανήκει ε, στο σιδηροδρομικό όμιλο της Κίνας και στις ουγγρικές σιδηροδρομικές γραμμές. Μία κοινοπραξία λοιπόν μεταξύ Ουγγαρίας και Κίνας. Τέλος πώς θα διασφαλίσουμε ότι θα ισχύσουν οι ε, κανόνες δημοσίων προμηθειών και πάλι δεν ήταν στο πεδίο ε, εφαρμογής της μελέτης μας. Ήταν μια τεχνική αξιολόγηση αυτή και εναπόκειται στα κράτη-μέλη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση να κρίνει κατά πόσο τηρήθηκαν οι κανόνες των δημοσίων προμηθειών. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίαση και για όλα τα στοιχεία που μας αναφέρατε. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον κύριο Πρέτη για αυτή τη μελέτη. Βρισκόμαστε μόλις στην αρχή νομίζω αυτής της συζήτησης και θα ασχοληθούμε περαιτέρω με αυτό το θέμα ως Επιτροπή Μεταφορών γιατί θα είναι μία από τις μεγαλύτερες προτεραιότητες ε, του μέλλοντος. Σας ευχαριστώ όπως και να έχει. Και συνάδελφοι, φτάνουμε στο τέλος της πρωινή συνεδρίασης. Παρακαλώ, κύριε Βαντερκάμπ. Πρόεδρε, θα ήθελα να επανέλθω στην πρόταση που έκανα και εγώ και ο Ισμαήλ Ερτούκ. Αυτή η μελέτη δηλαδή να εξεταστεί και στην αντιπροσωπεία για την Κίνα, στην αντιπροσωπεία για την Ασία, στην Ίντα ή στην ΑΦΕΤ. Ε, θα ήθελα παρακαλώ να το διαρευνήσετε πώς μπορεί να γίνει αυτό. Άκουσα με μεγάλη προσοχή τον κύριο Πρέτη. Ε, προσπαθεί να κρατήσει αποστάσεις του από τα γεωπολιτικά ζητήματα και το κατανοώ. Αλλά εμείς ως πολιτικοί έχουμε διαφορετικό καθήκον από ότι ένας ερευνητής. Ευχαριστούμε. Έχουμε σημειώσει την πρότασή σας. Γι' αυτό θα κάνω ό,τι μπορώ. Θα αποταθώ στις επιτροπές ΕΙΝΤΑ και ΑΦΕΤ προκειμένου μέσα στις επόμενες εβδομάδες να υπάρξει συντονισμός για να συζητήσουμε αυτό το θέμα, τον δρόμο του μεταξιού. Θα το εξετάσουμε λοιπόν και στην επόμενη συνεδρία των συντονιστών υπό ποια μορφή θα μπορέσουμε να εξετάσουμε αυτό το ζήτημα. Εντάξει. Ωραία, τα ξαναλέμε στις 2.30 και πάλι εδώ. Καλή όρεξη.